Uh, good morning, colleagues. Um, Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Άφησα να περάσει λίγη ώρα, μήπως και έρθει κανείς παραπάνω στην αίθουσα, εν πάση περιπτώσει. Καλή σας ημέρα. Και καλημέρα ιδιαίτερος και ευχαριστώ πολύ την κυρία Κάρνιετ, η οποία ως εισηγήτρια ήταν και παρούσα νωρίς νωρίς τη συνεδρίαση. Κφώματα. Θα κάνω κάποιες ανακοινώσεις αργότερα όμως. Κάποια θέματα που συζήτησαν οι συντονιστές, αλλά πρώτα θα ήθελα να περιμένω λίγο, μήπως έρθει κανείς ε, άλλος από τους συναδέλφου. Και γι' αυτό εντωμεταξύ θα προτείνω να προχωρήσουμε με την κυρία Κάλνιετε για την ε, γνωμοδότηση ως προς την ασφάλεια προμήθειας σε φυσικό αέριο που έχει συντάξει. Και μετά θα δώσω το λόγο στους Σκιώδη Μόνο ο κύριο Στρατεφλίδης είναι εδώ από ό,τι βλέπω από τους Σκιώδη, αλλά... Μέσα περιπτώσει. Ίσως και η κυρία Γκέμπχαρτ. α, ναι, και η κυρία Πέρμπαρτ. Κύριε Σίβιτσιτ. Δεν έχετε την ε, καρτέλα με το όνομα, γι' αυτό δεν σας είδα αμέσω. Έχετε καρτέλα αναπληρωματικού μέλους μπροστά σα, κύριε Σίβιτσι. Ναι, ευχαριστώ που με διορθώνετε για την προφορά του ονόματο. Επίσης, Έχουμε εκπρόσωπο τη ε, μονάδα ε, για την Ασφάλεια Προμήθειας Ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Κοντεσίβιτ από την ε, Μονάδα χάραξη πολιτική. Α, δεν είναι εδώ, μάλιστα. Θα μα μιλήσει μετά. Και αν είναι παρόν το Συμβούλιο, θα δούμε και τι δικέ του παρεμβάσει. Κυρία Κάλνιετε, λοιπόν, παρακαλώ. Με χαρά σα δίνω το λόγο να μα πείτε τι γνώμη έχετε για αυτή την πρόταση τη Επιτροπής. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξεκινώντας την παρουσίασή μου θα ήθελα να πω ότι θεωρώ σημαντικό να επικεντρωθούμε σε τέσσερα ζητήματα για τις ε, επιχειρήσεις φυσικού αερίου. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε την ε, προσπάθεια για εξασφάλιση των ε, προμηθειών σε ενέργεια σε επίπεδο αγοράς, υπηρεσιών και κοινοτήτων και Σε σχέση λοιπόν ε, και σε συνεργασία με τους ε, συναδέλφους και όδης συγητάς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η αρχή αυτή των τριών ε, επιπέδων δεν έχει διαρθρωθεί επαρκώς. Και υπάρχει ανάγκη να προσδοριστεί ο ρόλος και οι ευθύνε των επιχειρήσεων ως προς την αντιμετώπιση των κρίσεων. Μετά, έχω ασχοληθεί επίσης με το ζήτημα του προστατευόμενου καταναλωτού ή πελάτου. Προτείνουμε να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρμογής του όρου αυτού, προστατευόμενος πελάτης, ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική προστασία, ικανοποιητικές εγγύσεις. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει το πεδίο αυτό να είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη-μέλη διαφορετικά, θα έχουμε διαφορετικές, ε, διαφορετικές προδιαγραφές στα κράτη-μέλη με αποτέλεσμα εμπόδια και στις ε, ρυθμιστικές διατάξεις και στο κόστος αλλά και στην ε, αρχή της ελληνικής. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω την προτεραιότητα ως προς τους μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων. Μέτρα όπως αποθήκευση, αποχέτευση και άλλα μέτρα δεν μπορούν να αποκλειστούν ως μέτρα κατεπίκουσας ανάγκη σε περίπτωση κρίσεως. Αλλά αυτό μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέτρα που μπορεί να προτείνει η αγορά. Και εν τέλει, διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών σημαντικός παράγων. Οι συνάδελφοι και εγώ θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή απόψεων, ε, μηχανισμοί παρακολούθησης, ε, μηχανισμοί ενημέρωσης, αναφοράς και τι προτείνουμε για τα περαιτέρω. Προετοιμαζόμενοι για την έγκριση της γνωμοδότησης σε επίπεδο κοινοβουλευτική Επιτροπής τον Νοέμβριο, εγώ θα πρότεινα να ζητήσουμε περισσότερες διευκρινήσεις για αρκετά ζητήματα και καλό και τους σκιώδεις ηγητές ε, να συμμετάσχουν ε, στον αναλογισμό της υπόθεσης αυτής, καταρχάς ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί βλέπουμε ότι στην τροπολογία υπαριθμών 5 ίσως χρειάζονται περαιτέρω ε, ίσως χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία. Δεύτερον, ως προς την έννοια του προστατευόμενου πελάτου, διότι υπάρχουν πολλές αποκλίνουσες ε, ερμηνείε, γιατί κάποιοι θέλουν ο προστατευόμενο πελάτης να έχει, να έχει περιεχόμενο πολύ πιο ευρύ, λιγότερο αυστηρό. Ε, τρίτον, ανταλλαγή πληροφοριών ε, και εδώ τα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι διστάζουν, δεν προτιμούν να προσφέρουν πληροφορίες ως προς τις συμφωνίες οι οποίες καταλήγουν και ίσως θα ήταν καλό να πιέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως θα ήταν δυνατόν η ολοκληρωμένη συλλογή των πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών, ε, να, να γίνεται πρώτα ολοκληρωμένη συλλογή των πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών και μετά αυτά, αυτές να διαβιβάζονται στα κράτη-μέλη. Και επίσης ένα πακέτο για την ε, συνολική ρύθμιση της αγοράς ε, ενέργειας. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα συνολικά να πω ότι Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής. Καλώς ορίζουμε την πρόσκληση του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα για την υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο προτάσεων για τη θέσπιση μέτρων ε, για τους κατάλληλους και απαραίτητους μηχανισμούς. Όπως είπε το Συμβούλιο θα πρέπει οι ρυθμίσεις να υιοθετηθούν το ταχύτερο δυνατό και κατά την επεξεργασία αυτής της ε, γνωμοδότηση είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με εκπρόσωπου τη Επιτροπής και με όλους τους σχεδόν τους κοιόδους συγητάς και έλαβα υπόψη στο βαθμό που μπορούσα τις παρατηρήσεις όλων. Ως πρώην διπλωμάτης θεωρώ ακράδαντο ότι θα πρέπει και η Επιτροπή μας να έχει Λόγω στην υπόθεση αυτή και στις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις. Λόγω των ε, χρονικών όμως ε, πιέσεων επικεντρώθηκα μόνο στα κύρια θέματα, στα θέματα που θεώρησα ότι είναι πιο στενά συνδεδεμένα με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 11η Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι και προσκαλώ όλους τους χιώδης συγητάς σε συνεδρίαση στις 9 το πρωί, στις 11 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να αντιπαραβάλουμε τις θέσεις μας και να ε, προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα στην έγκριση νομοδότησης. Και παρακαλώ τους πάντες, εάν δεν είναι σε θέση, οι σκιώδεις ηγητές δηλαδή, εάν προσωπικός δεν είναι σε θέση ένας από εσάς να μην είναι παρόν, να δώσει πληρεξούς σε κάποιον άλλον συνάδελφο για να τον ε, αντικαταστήσει. Ε, και φυσικά δεν θα πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Επιτροπής μας για την υποστήριξη που προσέφερε, καθώς και όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Για το έργο σας και για όλη την προσφορά σας σε αυτή την Επιτροπή. Ακούσαμε την πρώτη σας σύλληψη του θέματος και το πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα σχετικά ζητήματα. Η γνωμοδότηση για αυτή την Επιτροπή λοιπόν είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά τους καταναλωτές, όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τα δικαιώματά τους βεβαίως. Είναι σημαντική λοιπόν η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και επιρροή στην εξέλιξη του όλου θέματος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερως. Τώρα, στον κατάλογο των αγορητών έχω τους κέντρους εισηγητές, τον κύριο Σίβιτ, τον κύριο Τρενταφυλλίδη. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να παρέμβουν. Ο κύριο Σμιτ, η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προχωρήσω κάπως περισσότερο στην κατεύθυνση που μας πέδειξε η συγγήτρια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε πολλές ε, συνομιλίες και διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και έχουμε ακούσει και τις απόψεις των ε, ενδιαφερομένων ομάδων καταναλωτών. και βεβαίω της ε, βιομηχανία παραγωγής φυσικού αερίου και διανομής αυτού. Ήταν λοιπόν η περίοδος αυτή μια περίοδος εντατικών εργασιών. Είχαμε τακτικές επαφέ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σαφώς γνωρίζουμε σήμερα πολύ περισσότερα για το θέμα. Αυτό από όταν ξεκινούσαμε. Γνωρίζουμε ποιο είναι το κοινό έδαφο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Υπάρχουν όμω τομεί. όπου υπάρχουν σαφεί διαφορέ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που και η συγγήτρια μόλις πέδειξε. Να σας πω, να σας θυμίσω ότι όταν πρωτοσυζητήσαμε το θέμα αυτό, καταλήξαμε εδώ ότι η έκθεση αυτή είναι σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, η παροχή φυσικού αερίου είναι σημαντική γιατί αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση και έπειτα Εάν δεν υπάρχει αξιόπιστη και σταθερή παροχή αερίου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό όπλο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, συνεχώς νέες απειλές που προκύπτουν από διαφορετικές πλευρές ε, στην αλυσίδα της παραγωγής και είναι ένα νέο στοιχείο αυτό, ένας νέος παράγοντας. Σκεφτείτε μάλιστα σε συνδυασμό με αυτή την απειλή και το στοιχείο της νέας γρήπης, την, το ενδεχόμενο πανδημίας. Λοιπόν, ο κίνδυνος που διαφαίνεται είναι σοβαρός. Τώρα πιο συγκεκριμένα για την πρόταση που εξετάζουμε. Έχω παρατηρήσεις ε, για δύο τροπολογίες συγκεκριμένα, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί και θα ήθελα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να επεξεργαζόμαστε αυτέ τι τροπολογίες. Για την τροπολογία υπαριθμών 3 προσπαθεί να διασφαλίσει καλύτερη προστασία για του καταναλωτέ η κατεύθυνση είναι ορθή αυτή που γενικώ ακολουθείται, αλλά δεν έχουμε κάνει αρκετέ προσπάθειες. Θα πρέπει να γίνει πιο σαφές και θα ήθελα να το επεξεργαστούμε περαιτέρω, διότι είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς ακριβώς θα δράσουμε σε αυτό το ζήτημα. Και για την πέμπτη τροπολογία, Στην τροπολογία παριθμών 5 η εισηγήτρια κάνει λόγο για πληροφόρηση για τις τιμές. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και πάλι, όμως δεν πηγαίνει αρκετά μακριά. Να περάσω τώρα σε πιο συγκεκριμένε παρατηρήσει, οι οποίε ελπίζω να πάρουν σάρκα και οστά σε συγκεκριμένε τροπολογίε, εφόσον καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει. Α δούμε το άρθρο 10, στο σημείο 1, όπου ορίζεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγεται ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να δηλώνεται ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός κράτη-μέλη. Όμως, μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης φαίνεται πιθανό και ενδεχόμενο να δηλώνεται και να αναφέρεται από ένα μόνο κράτος μέλος γιατί να μην φανταστούμε ότι μία χώρα θα έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα ζητήσει τη συνεργασία και τη συνδρομή άλλων κρατών μελών. Είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Μια άλλη μου παρατηρήση αφορά το άρθρο 7.5 στο σημείο 5 όπου αναφέρονται οι τιμές. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής διάκριση. Και εγώ πιστεύω στην αγορά και στην οικονομία της αγοράς και πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε την αγορά να λειτουργεί αυτόνομα και να ρυθμίζει μόνη τη τα θέματα τη στο βαθμό το δυνατού. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να προτείνω την εξή διατύπωση για το 7-5. Μετά την φράση που ήδη προτείνεται από την Επιτροπή, μετά τον όρο commodity, θα ήθελα να προσθεθεί το εξή. Θεωρώντα ότι η άσκηση τη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και υποχρεώσει για τι δημόσιε υπηρεσίε στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης επιβάλλουν τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την υπέρμετρη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Νομίζω ότι από αυτό διαφαίνεται ποια είναι η πρόθεσή μας. Δεν έχω λοιπόν περαιτέρω σχόλια. Τώρα, στην ίδια κατεύθυνση, ήθελα να προτείνω μια τροπολογία στο άρθρο 5D με την εξή διατύπωση. 5.1.D. Η πληροφόρηση και υποχρεώσει ε, δημοσίων υπηρεσιών καθώ και προστασία καταναλωτών όπω ορίζονται στην Οδηγία 3 τη Οδηγία 2001-23 καθώ και η λήψη μέτρων από τα κράτη-μέλη για την προστασία των καταναλωτών από την υπερβολική αύξηση των τιμών. Αυτές, κατά την άποψή μου, είναι τρεις σημαντικέ τροπολογίες και είναι σημαντικές για την πολιτική μου ομάδα. Θέλουμε να προστατεύσουμε εδώ τους ε, μεμονωμένου καταναλωτέ, τους ανθρώπους που διαβάζουν τις εφημερίδες, διαβάζουν τον τύπο και φοβούνται για την ασφάλεια της παροχή φυσικού αερίου. Ε, κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω κάποιε ε, μικρές αλλαγές, στο αρχικό τμήμα του κειμένου. Μια μαγική λέξη που ήθελα να αλλάξει και φαίνεται ότι είναι δύσκολο να την αναφέρουν κάποια κάτι μέλη, η αλληλεγγύη συγκεκριμένα. Δυσκολευόμαστε όλοι να αναφέρουμε την ε, αλληλεγγύη για να παραπέμπουμε σε αυτή, ιδίω περιπτώσεις περιπτώσει που υπάρχουν ε, μείζωνα προβλήματα για του πολίτε μα. Ο κανονισμός όμως σκοπό έχει ακριβώς αυτού να προστατεύει. Θα σεβαστώ βεβαίως απολύτως την ε, βούληση τη ε, συγγήτρια να ξανασυντηθούμε στις 11 του μήνα για να ξανασυζητήσουμε. Έτσι κι ε, σε μια εβδομάδα είναι η 11η του μήνα. Και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες αλλά θα ήθελα να ληφθούν υπόψη αυτές τις τροπολογίες που είναι η τοποθέτηση της πολιτικής μας ομάδας επί της ουσίας. Ο Πρόεδρος, κύριε Σιβίτσο, ευχαριστούμε και προσέξτε, η κυρία Κανέτη να λάβει εγκαίρω τι τροπολογίες σας. Ελήφθησαν υπόψη όσα είπατε, αλλά και εσείς να κάνετε αυτό που πρέπει να τις υποβάλλετε όπως πρέπει. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια τόσο για τη δουλειά της αλλά και για τη συνεργασία που είχαμε και θα εξακολουθήσουμε να έχουμε. Είχα μια συνάντηση με την εισηγήτρια στην οποία είχαμε εξηγήσει τη δική μας αντίληψη των πραγμάτων. Είχαμε πει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο για την διαχείριση των ενεργειακών του πόρων, ενός τομέα που αποτελεί σημαντικό οικονομικό άξονα για τα κράτη. Είχαμε επίσης πει ότι σε περιόδους έκτακτης ανάγκης θα πρέπει τα μέτρα που παίρνονται να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στην εκάστοτε κρίση. Βασικό δηλαδή κριτήριο δεν μπορεί να είναι ο βαθμός ανταπόκρισης στην εσωτερική αγορά, αλλά η αποτελεσματικότητα στη στήριξη των καταναλωτών. Αυτό το τελευταίο είναι που νομίζουμε ότι λείπει. Εμείς πιστεύουμε ότι η θέση ότι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που στηρίζεται αποκλειστικά στην εσωτερική αγορά, η οποία εκφράζεται ως βασική αρχή στον προτινόμενο κανονισμό, ότι αυτή η θέση θα επιλύσει το πρόβλημα εφοδιασμού είναι λαθασμένη. Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι η απουσία ελέγχου είναι γενεσιουργός αιτία των κρίσεων και μονομερός η αγορά δεν μπορεί να επιφέρει ασφάλεια στον εφοδιασμό. Ενώ η εισηγήτρια εγείρει το θέμα για προστασία των καταναλωτών, καμιά αναφορά δεν γίνεται για τον έλεγχο των τιμών και καμιά αναφορά δεν γίνεται για αντιστροφή της πλήρους απελευθέρωσης του τομέα της ενέργειας. Οι τροπολογίες 2 και 4 εισάγουν τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου ως φορέα στον οποίο θα κατανεμηθούν αρμοδιότητες για την υλοποίηση των διατάξεων του κανονισμού. Η εισαγωγή των επιχειρήσεων φυσικού αερίου συναρμόδιου φορέα με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την υλοποίηση των στόχων του κανονισμού δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών. Επομένως, εμείς κύριε Πρόεδρε θα καταθέσουμε τροπολογίες οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις αρχές που έχω εξηγήσει. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Σα ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα πάμε στου άλλου αδέλφου. Έχω εδώ εγγεγραμμένου. Σμιτ, Γκέμπχαρτ, Τσερκόφσκι και Ρότιμπαρ. Uh, Σμιτ, όχι. Ο κύριο Μάντερς είναι ο σκιώδη ηγητή. Σας εξηγώ απλώς γιατί, λαμβάνω τώρα το λόγο. Καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε, λέει ο πρόεδρος. Και ο κύριος Μπίλαν ε, επίσης παρίσταται, όπου είναι σχεδόν συγγητή. Οπότε φαντάζομαι και εκείνο θέλει το λόγο. Αν βλέπω, ξέρετε, τι θα πω πριν το πω. Πολύ καλό αυτό. Κάθε φορά κάνω μια ματιά σε κάποιο έγγραφο για το φυσικό αέριο ε, κάθε φορά θεωρώ ότι θα πρέπει κάθε φορά να ε, σκεφτόμαστε τι εναλλακτικέ πηγές ενέργειας υπάρχουν και άρα θα πρέπει να αναφέρουμε του, τους προς βοράν και προς νότο αγωγούς. Το Nord Stream, ας πούμε, που διέρχεται από την Βαλτική και κατά τη γνώμη μου υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα με το φυσικό αέριο και τον Nord Stream γιατί πρόκειται για αέριο. Ε, πρόκειται για εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακος. Ε, εκεί προέρχονται από τη Ρωσία. Και έχουμε εδώ ένα κείμενο το οποίο προτείνει κάποιες εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Δεν αρκεί το φυσικό αέριο. Πάντα θα υπάρχει πολιτική πίεση. παρά κάποιες τροπολογίες που εκφράζουν την αλληλεγγύη και βέβαια δεν μπορώ να διαφωνήσω θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ευρύτερα εμείς τουλάχιστον στην Επιτροπή μας γιατί θεωρώ ότι αν θέλει να δει τα πράγματα από πλευρά καταναλωτών θα πρέπει να τα δει κατά αυτόν τον τρόπο. η καρχιδόνα καταστράφει λέγανε και κάθε φορά λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία λέμε είναι διαπιστωτικά κάποιας, ε, ε κάποιας καταστροφής που θα έρθει. Επομένως, προσοχή, αυτό το θέμα δεν είναι, δεν είναι ρωσογερμανικό, είναι δικό μας. Α, πολύ ωραία, μας είπατε και λατινικά, Καρθάγκο Ντελέντα Εστ, λέει ο πρόεδρος και προχωρά. Ε, έχουμε εδώ νησιώδη συγκριτή τον κύριο Μπίλαν. Θέλετε το λόγο. Όχι, όχι, λέει ο κύριος Μπίλαν. Και ζητεί το λόγο η κυρία Γκέμπχαρτ. Α, ήρθε ο κύριος Μάντερς. Αλλά πρώτη ζήτησε το λόγο κυρία Γκέμπχαρτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, μας κάνετε πάντα να χαμογελούμε με το British humor που έχετε και πάντα μας διασκεδάζει στη δουλειά μας, περνάμε πιο ωραία. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο κυρία Κάλνιατε για τη δουλειά της, για τη συνεργασία και ευχαριστώ και τον κύριο Σίβιετς ε, που ως και εδώ δεν έχει την πλήρη υποστήριξη της ομάδας μου θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε να ε, ασχοληθούμε ως Επιτροπή και με την προστασία των καταναλωτών. Δεν μπορούμε να το λησμονούμε λοιπόν, λοιπόν αυτό. προστασία των καταναλωτών σημαίνει να μεριμνούμε εκεί ακριβώς που υπάρχουν ζητήματα προμήθειας ενέργειας και η προμήθεια σε φυσικό ε, αέριο είναι ενέργεια για ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδιαίτερες δυσκολίες και έχει τεράστια σημασία και εκεί πρέπει ακριβώς να δίνουμε και εμείς ιδιαίτερη έμφαση. Ως εκ τούτου οι τροπολογίες του κυρίου Σίβιετς είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, και κύριε Χάρμπορ δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στο εγκαίρως να υποβληθούν και να μπορέσει να τις ε, συμπεριλάβει η κυρία Κάλινετ στην ε, γνωμοδότησή της. Θα ήθελα να πω ότι η αρχή της οικουμενικής υπηρεσίας ε, στην ε, προμήθεια σε ενέργειες έχει τεράστια σημασία. Σημαίνει δηλαδή αυτή η αρχή ότι το κράτος φροντίζει, ελέγχει, επαληθεύει ότι παρέχεται η υπηρεσία που χρειάζεται, εν προκειμένου η προμήθεια σε φυσικό αέριο, για οποιονδήποτε τη χρειάζεται, την ώρα που την χρειάζεται, υπό τους όρους που τη χρειάζεται. Και εδώ ε, η έννοια του προστατευόμενου καταναλωτή για μας δεν είναι οι καταλληλότεροι γιατί είναι πολύ γενικόλογοι, εννοεί γενικά κάθε είδους καταναλωτή κτλ. Εμείς θέλουμε ιδιαίτερη έμφαση να δώσουμε στον πολίτη ο οποίος βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομικά κατάσταση, σε μια άλλου είδους ιδιαίτερη δυσκολία γιατί παραδείγματι είναι ε, ένα άτομο με αναπηρίες, γιατί έχει οικονομικά προβλήματα, γιατί είναι δύσκολη η πρόσβασή του στην προμήθεια σε φυσικό αέριο. Ε, όλα αυτά τα θέματα λοιπόν που αποτελούν για μας εταιρεία σημασία ζητήματα για την προστασία του καταναλωτή. Στην τροπολογία παριθμών 1 η αξιολόγησή μου είναι η ίδια με αυτή του κυρίου Σίβιετς. Σε προβληματικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε θέματα ε, νοικοκυριών, σχολείων, ε, νοσοκομείων θέλουμε ένα σαφή ορισμό των προτεραιοτήτων μας. Ποιος είναι πρώτος στη σειρά. Ενώ εσείς βλέπω ότι τα έχετε κάνει ένα συνονθήλευμα αναφερόμενο στη γενική προστασία του καταναλωτή. Πράγμα το οποίο οδηγεί σε αμφισβήτηση μέσω της τροπολογίας σας της προτεραιότητας που θα έπρεπε να δοθεί κατ' εμάς στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Πράγμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Γιατί το κάνετε αυτό. Τουλάχιστον να δω μια ε, εξήγηση λογική κάποια, ε, κάποια επιχειρηματολογία. Γιατί προβαίνετε σε αυτήν την επιλογή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκέπχαρτ. Ο κύριο Τρασκόφσκι, Μάντερς, ο σκιώδη εισηγητής για του ελεύθερου και κατόπιν κυρία Ρότεμπα. Κύριο Σκόφσκι. Τώρα το, το προφερώ όπως όπω το ονομάζα, λέει και τον άλλο κύριο Τρασκόφσκι. Από ό,τι φαίνεται Έχουμε κύριο συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά θα τεθεί σε ισχύ σε επόμενες μέρες. Οπότε για την Πολωνία και για άλλες χώρες θα πρέπει να τονιστεί ότι η αλληλεγγύη, τουλάχιστον για τα ενεργειακά θέματα, είναι κάτι που καλύπτονται συνθήκη κλπ. Άρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον κύριο Σίβιτς, ότι δηλαδή η λέξη αλληλεγγύη θα πρέπει να αναφέρεται στην ε, γνωμοδότηση. Να υπάρχει στο σώμα του κειμένου. Και θα πρέπει επομένω έτσι να ερμηνευτούν αυτά τα κείμενα, να ερμηνευτούν υπό το φω τη νέα συνθήκη. Άρα συμφωνώ με το να μπει η λέξη ελεγγύη στην γνωμοδότηση. Επίσης θέλω τώρα να συμφωνήσω με όσους είπαν ότι χρειάζεται να γνωμοδοτήσει η ΑΦΕΤ τόσο ώστε να επηρεάσουμε κάπω την εξωτερική πολιτική. Ακούσαμε τι είπε και ο κύριο Σμιτ για του αγού φυσικού αερίου και έτσι να δούμε το πώ θα αναφέρουμε κάτι και για ε, του αγού φυσικού αερίου. Βέβαια, ε, εμεί ασχολούμαστε με την εξωτερική αγορά και επομένω είναι κυρίω δουλειά τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να αποφανθεί για αυτά τα ζητήματα. Τρίτον. Η κυρία Κανιέτε επετέλεσε πάρα πολύ στο έργο και συμφωνώ με τους κυρίους Σίβιτς και την κυρία Κέμπχαρτ αλλά δεν καταλαβαίνω τι, τι έγινε με την ε, τροπολογία που ε, αναφέρθηκε την παρθμόν 1. Τέλος. Για την ανταλλαγή πληροφοριών θέλω να σας πω. Όσον αφορά αυτή την προπόθεση του να υποβάλουν τα κράτη-μέλη όλες τις συμφωνίες με τρίτε χώρες που έχουν επίδραση στις ε, υποδομές και τα δίκτυα παροχή του φυσικού αερίου Επίση απαιτείται τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε την διατύπωση, να την κάνουμε κάπως πιο αυστηρή, πιο δυναμική. Γιατί εκεί που λέει για την επίδραση στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Ποιος θα κρίνει ποια συμφωνία έχει κάποια επίδραση. Φοβάμαι ότι τα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να κοινοποιήσουν αυτές τις συμφωνίες στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχυριστούν ότι η συμφωνία που συνήψαν δεν έχει επιρροή στη, στο φυσικό αέριο. Ε, το ίδιο ισχύει και για, για την συμμόρφωση προς την νομοθεσία. Άρα να γίνει διατύπωση κάπως πιο δυναμική, να γίνει αυτό κάπως πιο δεσμευτικό. Πάμε να το κοιτάξουμε πώς υποβάλλω και η τροπολογία. Άρα, συμφωνώ με τους συναδέλφους και σας επισημαίνω τα της αλλαγής της διατύπωσης, τόσο ώστε να γίνει πιο δεσμευτική διατύπωση. Harbor. Πάρα πολύ θετικά όσα μας είπατε και δίνει το λόγο στον κύριο Μάντερς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνάδελφη κυρία Κάρνιετε για την ε, συνεργασία. Έχουμε ήδη συζητήσει για το θέμα αυτό πολλές φορές. Για τον κανονισμό διερωτώμε εάν υπάρχει δυνατότητα να τεθεί σε ισχύ πριν ε, πιθανότητα μάλλον το θέσει ισχύει πριν από την οδηγία για το φυσικό αέριο που υιοθετήσαμε πέρυσι και ακόμη δεν έχει αρχίσει να εφαρμόστε επειδή δεν την έχουν θέσει εφαρμογή τα κράτη-μέλη. Ερωτώ λοιπόν εάν μπορούμε να ελπίζουμε στην εφαρμογή της περίπου ε, δύο εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του κανονισμού. Θα πρέπει εντωμεταξύ να διαφωνήσω λίγο με τον συνάδελφο Όλε για τους ε, αγωγούς ε, όπου θεωρώ ότι θα έπρεπε το εγχείρημα για, τους, για τον αγωγό φυσικού αερίου να μην είναι μόνο ρώσο-γερμανικό, αλλά ευρωπαϊκό επιχείρημα, ευρωπαϊκή επιχείρηση. Ίσως θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε αυτό με κάποια τροπολογία. Είχαμε προτείνει να υπάρχει μια σύνδεση όλων των κρατών μελών μέσα από την Ήτρε πέρυσι. Μέσα από ε, την Ήτρε λοιπόν είχαμε προτείνει να υπάρχει σύνδεση όλων των κρατών μελών στο σύστημα για το φυσικό αέριο, για την εξασφάλιση της προμήθειας σε αέριο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει κανένα κράτος να βρεθεί αποκλεισμένο. Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται και η φυσική μεταφορά του αερίου. Είναι πολύ δύσκολο το να λάβει αυτό ένα κράτος μέλος μόνο του και ίσως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη αυτή της ανάπτυξης ενός δικτύου φυσικού αερίου ε, στην Ευρώπη, πέραν των συνόρων. ώστε να μπορεί ο κάθε καταναλωτής να έχει εγγυημένη την προμήθεια σε αέριο. Ω προ το κείμενο θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά σημεία κοινά. Θα έλεγα ότι είναι αντίγραφο των όσων θετήσαμε πέρυσι με την ε, πρόταση οδηγία. Αν και σημειώνω εγώ ότι πάντα προτιμώ του κανονισμού και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κανονισμό ε, και άρα μπορούμε να περιμένουμε ταχύτερη εφαρμογή του σε σχέση με την οδηγία. Ίσως μπορούν ε, οι νομικές, η νομική υπηρεσία να μας ενημερώσει και να μας εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτή η στρέβλωση στο δίκαιο, δηλαδή γιατί δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία. Και ερχόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κείμενο, ίδιο κείμενο σωστικά στον κανονισμό αυτων Γιατί λοιπόν αυτή η στρεβλή κατάσταση στο δίκαιο. Ελπίζω να μας δώσει κάποιος μια ικανοποιητική απάντηση. Και τα άλλα, πιστεύω ότι θα είναι καλή και ισορροπημένη πρόταση και ελπίζω να την υιοθετήσουμε σύντομα. Um, Η κυρία Ρόιτοβα και ο κύριος Σίβιτς. Μπορείτε να δευτερολογήσετε. Και μετά εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτά όλα τα οποία έγιναν ε, πέρσι σε σχέση με το φυσικό αέριο μας ε, άγουν ίστο ε, να θέλουμε να διεκπαιρεωθεί αυτό το κείμενο όσο γίνεται γρηγορότερα. Και συμφωνώ με τον κύριο Μάντερς ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Τώρα, θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, διότι πάρα πολύ σωστά έχουν συνεργαστεί οι συγητές, οι σκιώδες συγητές και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις τροπολογίες. Όσον αφορά τον κανονισμό, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει το Συμβούλιο και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε μήπως επιβαρύνουμε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Μήπως θα ήταν επομένως καλύτερα να το διατυπώσουμε κάπως αλλιώς, να πούμε δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη θα δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις που εμπορεύουν το φυσικό αέριο κλπ. κλπ, κλπ. Να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους διατύπωση. Όπως το κάνουμε άλλωστε σε διάφορα νομοθετικά κείμενα.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 Δηλαδή 11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 διέπει τον κανονισμό αυτό και προέκυψε από την κρίση του φυσικού αερίου τον Ιανουάριο. Ότι θέλουμε να οικοδομήσουμε μια εσωτερική αγορά, διότι η εσωτερική αγορά είναι ο μόνο τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ροέ αερίου που να πηγαίνουν από δυτικά προ Ανατολά και ε, αντιστρόφω και από βορρά προ Νότο και αντιστρόφω. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλι το αέριο μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευρωπαϊκό και δεν πρέπει να σταματά να ρέει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεμπόδιστο. Αυτό είναι το πλεονέκτημα τη εσωτερική αγορά και αυτό είναι ο στόχο μα. Το μόνο φραγμό που απομένει εδώ και μπορεί να προκύψει είναι η έλλειψη υποδομών. Εκεί πρέπει να χτίσουμε τι απαραίτητε υποδομέ που μπορούν να περάσουν το αέριο από τα δυτικά προ τα ανατολικά. Αυτό χρειάστηκε να γίνει τον Ιανουάριο, αλλά ακριβώ γιατί είχαμε διακοπή από ανατολά προ δυτικά μπορεί να χρειαστεί. Λοιπόν, να ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να επιληθούν και αυτά τα προβλήματα των υποδομών θα εξετάσει ο ερχόμενο ε, κανονισμό. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν τα κίνητρα για να χτιστούν οι απαραίτητε υποδομέ, να λειτουργήσει εύρυθμα η εσωτερική αγορά και να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση και ασφάλεια στην παροχή φυσικού αερίου. Οπότε είναι πολύ σημαντική η αγορά. Δεν θα πρέπει να ιτηθούμε από μέτρα τα οποία μονομερώς λαμβάνονται από κράτη-μέλη. Αυτό αντι στρατεύεται την αρχή της αλληλεγγύης και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη των τιμών, διότι η αγορά εξελίσσεται και τα σημάδια που περιλαμβάνουμε, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις τιμές είναι σημαντικά. Δεν θέλουμε λοιπόν διωγγωμένες τιμές, αλλά θέλουμε τιμές που να πληρώνουν την ασφάλεια της παροχής. Δηλαδή, σε περίπτωση έλλειψης αερίου θα πρέπει να ανέβει τιμή λογικά του προϊόντος για περιορισμένο χρονικό διάστημα ενδεχομένω, αλλά σε αιτήσια βάση η τιμή μπορεί να παραμένει σε λογικά επίπεδα. Εάν δείτε τι έγινε όμως τον Ιανουάριο, επί δύο εβδομάδες υπήρχε έλλειψη αερίου και ήταν ξεκάθαρο ότι αν έπρεπε να πληρώσει κανείς επί δύο εβδομάδες περισσότερα τον αέριο, στο καταχύμωνο, ήταν το τίμημα που έπρεπε να καταβάλουμε για να έχουμε την ασφάλεια της παροχή. Βέβαια δεν πρέπει να πατούμε από τον φορολογούμενο να πληρώνει τη διαφορά ή... Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικός ο ορισμός των προστατευόμενων καταναλωτών, πελατών. Θα πρέπει πάντω να προσέξουμε να μην διευρύνουμε τον ορισμό αυτό καλύπτοντα όλου του πελάτε του αερίου. Δεν μπορεί ο μικρό φορολογούμενο να πληρώνει και να μην πληρώνει μεγάλε εταιρείε. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να έχουμε και τη δυνατότητα να περάσουμε Υπάρχουν μάλλον μεγάλοι πελάτε που έχουν τη δυνατότητα να περάσουν από το αέριο σε κάτι άλλο. Αυτοί οι προστατευμένοι λοιπόν πρέπει να μα απασχολήσουν. Διότι αν τη διευρύνουμε την έννοια και καλύψουμε μικρομεσαίε επιχειρήσει και άλλου, θα αυξήσουμε και άλλο την τιμή την ίδια διωγγωμένη προκειμένου να προστατευτούν και αυτοί οι πελάτες. Υπάρχει λοιπόν σαφή σχετισμός μεταξύ της έκτασης της έννοιας αυτής των προστατευμένων πελατών και του τιμήματος που θα πρέπει να καταβάλουμε. Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις. Και αναμένουμε διακαώσεις τις τροπολογίες σας θα είναι μια καθοριστική συμβολή στην όλη συζήτηση. Βεβαίω, η βασική καθήλυνα αρμόδια επιτροπή εδώ είναι η Επιτροπή Ήτρε. Θα έχουμε λοιπόν, νομίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση και εκεί, αλλά οι τροπολογίε που σημειώσαμε είναι μια χρήσιμη συμβολή στην όλη συζήτηση. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάλινετε για να κάνει την συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων της. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς όλους τους συναδέλφους. Ήταν ε, πολύ χρήσιμη η συζήτηση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να την αναπτύξουμε κατά τρόπο επικοδομητικό με όλους τους και οδησηγητάς για να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα υποβάλουμε προς έγκριση στις αρχές Δεκεμβρίου για να υιοθετηθεί από την Επιτροπή μας. Επίσης, για όσους δεν ήταν παρόντες την ώρα που παρουσίαζα το κείμενό μου, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχουμε την 11η Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Καλό δε όλους τους και ηγητάς σε συνεδρίαση στις 9 το πρωί, την ίδια ημέρα 11 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να συγκρίνουμε να αντιπαραβάλουμε τις θέσεις μας και να προχωρήσουμε απρόσκοπτα στην διατύπωση μιας κοινής, ε, ενός κοινού κειμένου και τη γνωμοδότηση ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την πρότασή μας το χειρότερο δυνατό. Από εκεί και πέρα ε, ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι εξής, όπως είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Όσον αφορά το, τα δικαιώματα του καταναλωτού, αντιλαμβανόμεθα ότι ίσως χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία η πρόταση και περιμένω προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους κοιοδησηγητάς. Δεύτερον, η έννοια του προστατευόμενου πελάτη είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Υπάρχουν τάσεις αυτών που θέλουν να διευρύνουν το πεδίο του ορισμού ενώ εμεί πιστεύουμε ότι αν διευρυνθεί το πεδίο του ορισμού θα καταλήξουμε σε έναν ορισμό ο οποίο θα καλύπτει του πάντε και ω εκ τούτου δεν θα είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν εγγυήσει για, για την προμήθεια σε φυσικό αέριο εκείνων που όντω το χρειάζονται. Σημαντικό λοιπόν για μένα είναι το γεγονός ότι αυτός ο ορισμός δεν ε, διαφέρει δεν θα διαφέρει ως προς την ε, εφαρμογή του ε, μεταξύ των κρατών μελών. Θα έχει δηλαδή, ε, θα εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο από όλα και σε όλα τα κράτη-μέλη. Ως προς την ενημέρωση, τη σχετική με τις διεθνεί συμφωνίες που συνάπτει ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική θέση, διαφορετικέ θέσει. Γι' αυτό και πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε πόσο θα βρούμε μια πολύ καλή λύση. Και επειδή και όπως το προσδιορίσαν και οι συνάδελφοι υπάρχουν οι προτάσεις αυτές οι οποίες σχετίζονται με την συνοχή του κανονισμού καθώς ε, ξέρουμε ότι έχει αποκλειστεί η Λετωνία από, την, ε, από το North Stream. Εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρόταβα και τον κύριο Σμίτ για την υποστήριξη που προσφέρουν, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνουμε και ότι, έχουμε να κάνουμε μια ιστορική, ότι είμαστε μια επιτροπή εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών. Και ο κανονισμός δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική διακήρυξη, διακήρυξη θέσεων. Και γι' αυτό οι τροπολογίες μας θα πρέπει να καλύπτουν θέματα των αρμοδιοτήτων μας και να μην ξεφεύγουν από αυτά. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου προσφέρατε και το αίτημα να συμπεριληφθεί ως θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ως διμερές θέμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, λέει ο ομιλήτρια, θέμα. Μα είναι και ηλίθεια μεταξύ άλλων. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Και... Πριν προχωρήσουμε στην ε, έκθεση της κυρίας Τσούν, θα ήθελα να κάνω τις ανακοινώσεις μου για τις ε, αποφάσεις των συντονιστών. Ελπίζω ότι θα το προσέξατε, ότι οι συντονιστές έχουν μια νέα πολιτική. Να σας ε, γνωστοποιούμε όσο γίνεται πιο νωρίς, αμέσως αφού συναντηθούμε, ένα χαρτί που θα λέει τι συζητήσαμε. Αλλά δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τους συντονιστές διότι συνεργάστηκα μαζί μου και έτσι βοηθούν το να δούμε τι θα γίνει με τις ε, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, με κάποιες ακροάσεις, με κάποιες μελέτες και τα πιο σημαντικά σημεία από τις χθεσινές συζητήσει, όλα αυτά τα αναφέρουμε εδώ και λέμε ότι έχουμε δώσει τέσσερις εκθέσεις σε τέσσερις συζητητές. Για τέσσερις εκθέσεις οικονομοθετήσεις. Πρώτα πρώτα, απαλλαγή προπολογισμού. Ε, θα το κάνει αυτό το ΕΛΚ. Επίσης, εφαρμογή του δικαίου πνευματική ιδιοκτησίας. Άλλη. Πολιτική ανταγωνισμού. PCR. Άλλη. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική αναφορά όσον αφορά του κάποιους ε, κανόνες για την άσκηση ε, της φαρμακευτικής πολιτικής, της πολιτικής περί στην Ισπανία και προσέξτε Έχουμε προτείνει και αντιπροσωπείε για αποστολέ σε άλλε χώρες. Ισπανία, Ινδία και σε κάποια χώρα του ε, Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Ελβετία ή Ισλανδία, οι μέρες δεν τις ξέρουν, θα σα τις πούμε. Επίση, συζητήσαμε και τα των ακροάσεων των υποψηφίων επιτρόπων. μόλι ξέρουμε τι θα γίνει, θα σας πούμε ποιες είναι οι ημερομηνίες. Επίσης, για τις ακροάσεις συζητήσαμε για κάποια εργαστήρια, για κάποια ενημερωτικά σημειώματα επίσης. Σημειώστε την 17η Δεκεμβρίου. Τελευταία Πέμπτη πριν τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές. Όσον αφορά το Συμβουλίο Ανταγωνιστικότητας, η Σουηδική Προεδρία ε, ήθελε να μας μιλήσει και η κυρία Σαμπούνι και Μπιούλιν ε, θέλησαν να έχουν μια τηλεσυνεδρίαση μεταξύ 10 και 12 στις 17 Δεκεμβρίου το πρωί. Οπότε παρακαλώ όσοι θέλετε ελάτε, όσο είναι πιο πολύ. Επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έντεση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Ζήτησε τηλεσυνεδρίαση μαζί μας όσον αφορά την οδηγία, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τώρα αυτό που προσπαθούμε να δούμε πώς προς τεχνολογίες αυτό θα υποστηριχθεί. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε τεχνολογία που έχουμε, μέσω της οποίας με βλέπετε και τώρα, σε οθόνη, αν θα μπορέσουμε λέγω έτσι να έρθουμε σε επαφή με την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Αυτά όσον αφορά το τι αποφάσισαν οι συντονιστές. Κάτι άλλο πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε σαν θέμα τώρα την επιτροπολογία δηλαδή. Κατά πόσον θα υπάρχει κάποια ανάθεση αρμοδιοτήτων μέσω της οποίας θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις η EFD, η ομάδα ήθελαν να συζητηθεί αυτό χτες όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς όπου έχουμε κάποια κατόφλια για την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας. Υπάρχει και διεθνή συμφωνία ο, και σύμφωνα με το κατόφλι το οποίο ισχύει θα πρέπει να γίνεται μια τακτή, η τακτική προσαρμογή. Και αυτό, αυτό έχει να κάνει με τα ειδικά τραβητικά δικαιώματα που προβλέπονται από τις διεθνείς συμφωνίες. Από το 1990 ξεκίνησε αυτή η ιστορία, έχει γίνει αναπροσαρμογή 12 φορές, αλλά τώρα κατεβάζει καινούργιες προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προσαρμοστούν αυτά τα κατόφλια και οι συντονιστές είπαν ότι δεν θα πρέπει να ε, έχουμε αντίρρηση όσον αφορά αυτό το μέτρο. Κάτι από αυτού. Ευχαριστώ απλώς να θυμίσω την ε, έκκληση του κυρίου Μέσα Σμιτ να ψηφίσουμε ως απάντηση για τα κριτήρια υπολογισμού και την αξιολόγηση της εκτιμήσεις για την αύξηση των τιμών στις στα διάφορα νομίσματα. Τον πίνακα που μας παρουσιάστηκε χθες δηλαδή με την αύξηση του 6% όπως χθες ζητήθηκε και υπόθηκε. Δεν καταλάβαμε ακριβώ πώ έγινε ο υπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σημείο προ σημείο την ε, μεθοδολογία που ακολουθήθηκε πριν μπορέσουμε να περάσουμε σε μια ψηφοφορία. Όχι, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, και ο Πρόεδρος. Είπαμε επομένω να μην ε, υποβάλουμε κάποια ένσταση όσον αφορά αυτή την πρόταση. Και είπαμε να ζητήσουμε να μας δώσει τον τρόπο, τη μέθοδο υπολογισμού η Κομισιόν που χρησιμοποίησε. Και είπαμε να έχουμε όχι μόνο σε ευρώ, αλλά και σε άλλα νομίσματα τα σχετικά ποσά των κατοφλίων. Και όσον αφορά βασίλειο, το κατόφλι ανέβηκε λόγω αλλαγής των τιμιών. Συμφωνείτε ωραία. Σημειώνω. Και έχω μια τελευταία ανακοίνωση. Χθε βράδυ πήγα στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής που αφορούσε την τελική φάση διεκπαιρέωσης του πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες ε, από πλευράς ε, Επιτροπής Βιομηχανίας συμμετείχε το Κοινοβούλιο και πάρα πολλοί από έχετε ασχοληθεί με αυτό, έχετε ασχοληθεί και με ε, τα καθολικά δικαιώματα και υπηρεσίες. Τώρα είναι ένα κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Είναι νομίζω θέμα δικό μας και θέμα το οποίο είναι μεγάλο επίδειγμα για τους καταναλωτές όλες οι πολιτικές πτέρυγες του Κοινοβουλίου ομόφωνα συμφώνησαν. Συμφωνήσαμε να γίνει μια τροπολογία. Ούτως ώστε να κατοχυρώνουν τα δύο σε κάποιες δύσκολες ε, περιπτώσεις όπου ίσως έχουμε κάποια αποσύνδεση από το διαδίκτυο ε, όπως ας πούμε κατάχρηση του copyright και συμφωνεί με το Συμβούλιο να υπάρξουν εγγυήσει για διαδικασία αμερόληπτη και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του θυγωμένου. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με τις προτάσεις μας και θα υπερψηφίσετε ό,τι τεθεί σε ψηφοφορία στην ε, ολομένη την επόμενη εβδομάδα. Εγώ συμμετέσχω σαν πρόεδρος Επιτροπής και σαν μέλος της, ε, της πολιτικής μου ομάδας. Μία η ώρα, μία το τα τελειώσαμε, οπότε συγχωρήστε αν είμαι λίγο κουρασμένος. <laughs> Uh, uh, let's move on. Uh, Mrs. Turnen Holstein, uh, uh, again, uh, thank you very much for the work you're doing for your first report for this committee. Um... Κυρία Τούν, Χόινστάιν, έχει τρώει το λόγο. Ευχαριστούμε για το έργο που επιτελέσατε. Έχουμε και τους ε, σκιώδους ηγητές, Γκέμπχαρτ, Ρούλε, Μπίλαν. Είναι οι σκιώδους ηγητές που παρίστανται. Κύριε Τούν, έχετε το λόγο. Ε, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak, to jest rzeczywiście mój pierwszy raport, bo niedawno Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι όντω η πρώτη μου έκθεση νεοεκλεγέν μέλος. Και στα θέματα του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς ήθελα να πω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ε, έχουμε μια περίοδο ενημέρωσης, την οποία καταγράφει, σχετική με την εφαρμογή ή καλύτερα την μεταφορά σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό δίκαιο των οδηγιών, αν και είναι ένας όρος που δεν προτιμώ να χρησιμοποιώ. Αυτός ο πίνακας λοιπόν αποτελεσμάτων ουσιαστικά καταγράφει την ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να φτάσει σε ένα ποσοστό 1% το οποίο αντιστοιχεί σε έλλειμμα μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εμεί φυσικά έχουμε διατηρήσει τον ίδιο στόχο, αλλά δεν βλέπουμε πώ θα τον επιτύχουμε το στόχο αυτό όταν 6% των οδηγιών δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι στόχοι λοιπόν τη καταγραφή αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων δεν είναι μόνο να έχουμε μια σαφή, καθαρή, αποτελεσματική, διαφανή εικόνα της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή της μεταφοράς των οδηγιών στις ε, εθνικές νομοθεσίες, αλλά και να επισημάνουμε ε, τι είδους προκλήσεις έχουμε μπροστά μας και τι είδους ευκαιρίες πρέπει να δράξουμε εγκαίρως. Εδώ μιλώ και για τις οδηγίες που δεν έχουν θέσει εφαρμογή τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για, τα, για την νομοθεσία που βρίσκεται στο τελευταίο κομμάτι του πίνακα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πίνακο εκ τούτου είναι ένα καλό μέσο να ασκηθεί πίεση προ τα κράτη-μέλη και τι κυβερνήσει του, ώστε ταυτόχρονα και να ευαισθητοποιηθούν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορεί ώστε να βελτιωθεί στο βαθμό του δυνατού η εσωτερική αγορά, γιατί πρέπει να βελτιωθεί. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, κάποιες τροποποίησεις για τους επόμενους. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τους επόμενους πίνακες. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με λεπτομέρειε ω προ την ε, μεταφορά σε εθνικό δίκαιο των ε, οδηγιών από τη συζητήση μου και μου το είπε άλλωστε ξεκάθαρα και η Επιτροπή, βλέπω ότι το έγγραφο αυτό είναι σαφές και αρκετά συνοπτικό ώστε να έχει την απαιτούμενη διαφάνεια. Αν προσθεθούν και άλλες πληροφορίες μέσα θα ε, είναι ο όγκος του τέτοιου μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, εγώ προτείνω να ε, ανοίξει μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ που θα μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο πολίτης ή όποιος ενδιαφερόμενος, να έχει τις λεπτομέρειες φερρυπίν από την ώρα της έγκρισης οδηγίας μέχρι την ώρα της θέσης εφαρμογής στο κάθε κράτος μέλος κτλ. Η ιστοσελίδα στο ίντερνετ δεν έχει τους περιορισμούς που έχει ε, το έγγραφο και γι' αυτό την προτιμώ. Επίσης, το Single Market Assistance Services, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει υποβάλει διάφορα σχέδια και προτείνω αυτά να υπαχθούν σε μια άλλη ιστοσελίδα στο ίντερνετ που να δίνουν ε, τα στοιχεία για τον πολίτη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, για τις επιχειρήσεις. Όπως δηλαδή χρειάζεται ο καθένα τα στοιχεία αυτά ε, για την ε, συμμετοχή του στην ιστορική αγορά και για την απρόσκοπτη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Αγορά. Υπάρχουν δύο πίνακε αποτελεσμάτων τη Επιτροπής. Ένας δύο φορέ τον χρόνο και άλλος ένας ετήσιος αυτή φορά που αφορά τον καταναλωτή. Η πρότασή μου λοιπόν είναι η εξή. Να συντονιστεί καλύτερα ο χρονισμός αυτών των πινάκων και έτσι να παρουσιάζονται, να δημοσιεύονται ταυτόχρονα. Και εγώ θα πρότεινα επίσης να έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε τα θέματα αυτά ταυτόχρονα. Και ταυτόχρονα εμεί, εφόσον υπήρχε αυτή η ταυτόχρονα δημοσίευση, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια διάσκεψη με συμμετοχή εκπρόσωπων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε αυτό που θα ονόμαζα εγώ το Φόρουμ Εσωτερική Αγορά να είχε την ευκαιρία να συζητά τα θέματα αυτά, τα προβλήματα ενδεχομένω που υπάρχουν, να προβάλλει τις βέλτιστες πρακτικές και να λαμβάνει και νέε δεσμεύσει ω προ την πιο αποτελεσματική οίθεση εφαρμογή των οδηγιών στα κράτη-μέλη. Θα ήταν καλό να έχουμε δέσμευση από τα κράτη-μέλη, όχι μόνο από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και η Επιτροπή των Περιφερειών, η Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή. Θα πρέπει να, συμμετάσχουν, να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο φόρουμ ε, για να υπάρχει μια πιο καλή εικόνα της εσωτερικής αγοράς, του τρόπου λειτουργίας, της, της ε, εφαρμογής των οδηγιών και της συμβολής στη λειτουργία της αγοράς. Διότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι ένα από τα πιο λαμπρά σημεία του ευρωπαϊκού ε, οικοδομήματος. Σε αυτό θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και να μεριμνήσουμε ώστε να εφαρμόζονται όντω οι οδηγίες τη εσωτερική αγορά και να φροντίσουμε η ε, δική μας πίεση να παραμείνει ε, και η παρουσία μας να παραμείνει ισχυρή για να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή. Εγώ ως νέο μέλος ομολογώ ότι ε, ανέπτυξα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καταρχάς το κείμενο, αλλά πάνω απ' όλα της, ε, τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και συναδέλφους. Πολλά στοιχεία ε, καινούρια έμαθα, συνεργάστηκα με τους κοιόδης με την Επιτροπή, με τη Γραμματεία της Επιτροπής μας, με τον κύριο Πετρούτσι που είναι εδώ, τον κύριο Κλενόφσκι, και ελπίζω ότι στο μέλλον θα γίνεται τακτική ε, δημοσίευση των ε, πινάκων αποτελεσμάτων με βάση τις υπόλοιπες προτάσεις τις οποίες έχω υποβάλει έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε κατά τρόπο συστηματικό τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Uh, uh, σας ευχαριστούμε κυρία Τούν ε, για τις συναρπαστικές αυτές πληροφορίες που μας δώσατε και τις ενδιαφέρουσες ιδέες σας. Ο καθηγητής Μόντι Διορίστηκε άλλωστε από τον πρόεδρο της Επιτροπής να ηγηθεί ειδική έρευνα στην επαναθέρμανση τη εσωτερική αγορά και την όλη διαδικασία. Οι συνάδελφοι λοιπόν θα παρακολουθήσουν και θα συνδράμουν στην προσπάθεια του τον καθηγητά Μόντι. Είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να συναντήσει μέλη της Επιτροπής λοιπόν και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το διοργανώσουμε αυτό, αλλά Ακριβώς η έκθεση αυτή θα συναρμοστεί αρμονικότατα με τη δική του τη μελέτη. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Γκέπχαρτ. Θα ακούσουμε και τους σκιώδεις εξηγητές, τον κύριο Σφάπ δηλαδή. Άλλος κανείς. Ωραία, αρχίζουμε με την κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ που είπατε και εσείς για άλλη μια φορά ότι ο κύριος Μόντι απεδέχθη τα σημαντικά αυτά καθήκοντα και ότι έχουμε υποσχεθεί ε, μέσα από μια έκθεση πρωτοβουλίας να παρακολουθήσουμε την υπόθεση αυτή και όχι μόνο σε σχέση με την ε, με μονομένη αυτή η έκθεση που αφορά του ε, πίνακε αποτελεσμάτων, αλλά με μια γενικότερη έκθεση πρωτοβουλία. Εγώ δεν είμαι σκιώδη ηγετρία τη ομάδα μου, πλην όμω ο κύριο Λίμουαν Κοκ, ε, συνάδελφο, δυστυχώ λόγω τη απεργία στο Ταλί, στου γαλλικού συντηροδρόμου, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα και γι' αυτό. Από ό,τι φαίνεται και η κυρία Βερνιό, η άλλη συνάδελφο δεν μπόρεσε να έρθει. μάς περιπτώσει μου έδωσε το κείμενό του στα γαλλικά και είμαι υποχρεωμένη να το αναγνώσω. Είναι το πιο εύκολο αυτό και στη συνέχεια θα ε, κάνω και τα προσωπικά μου σχόλια βέβαια. Αλλά τώρα διαβάζω στα γαλλικά για τους ε, για τους διερμηνείς. Ο κύριος Βουανκόκ που είναι σκιώδης συγγητής, παρακαλεί να συγχωρήσετε την απουσία του. Ε, χρειάστηκε να φύγει νωρίτερα, εχθές δηλαδή, λόγω της προβλεπόμενης για σήμερα απεργίας των Ταλής και μου δίνει εξ ονοματός του το σχετικό κείμενο. Ο κύριος ε, καταρχάς ευχαριστεί την συγγήτρια κυρία Τούν για την ποιότητα της ε, έκθεσής της και για την διάθεση για συνεργασία με τους σκιώδης συγγητάς. Όπως είπε και η συγγήτρια, μπορούμε να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και το γεγονό ότι ύστερα από ε, τον τρίτο αυτόν πίνακα αποτελεσμάτων τη εφαρμογή των ε, ε, οδηγιών παραμένουμε σε επίπεδο χαμηλότερο του 1% από αυτό που είχαν προσδιορίσει αρχή κρατών και κυβερνήσεων το 2007. Πλην όμως υπάρχουν νέα κράτη τα οποία δεν έχουν αρκετά καλό, καλά αποτελέσματα στη μεταφορά των οδηγιών και υπάρχουν ακόμη αρκετά τα οποία δεν έχουν θέσει εφαρμογή οδηγία, τη οποία η προθεσμία ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο έχει λήξει εδώ και δύο χρόνια. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα προβλήματα και πέραν αυτών των οδηγιών υπάρχουν και προβλήματα ω προ την, την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών, δηλαδή δεν έχουν σωστά εφαρμοστεί οι οδηγίε και άρα τα αποτελέσματα, τα ποσοστά δεν είναι το 1% που είχαν προβλέψει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά 8% και έτσι η Γαλλία, και ειδικότερα για να αφαιρθούμε στη Γαλλία, η Γαλλία έχει πολύ καλά αποτελέσματα με 0,8%, δηλαδή 13 οδηγίε που δεν έχουν ε, εφαρμοστεί, είναι 7η από τα 27 κράτη-μέλη, αλλά πέραν τη έγκαιρη θέση εφαρμογή έχει πρόβλημα στην ορθή εφαρμογή περισσότερο, ε, δηλαδή δεν, γίνονται, δεν γίνεται σωστά η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του περιεχομένου των οδηγιών και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν προσπάθειε έτσι ώστε όχι μόνο, εγκαίρω αλλά και ορθά να γίνεται μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών, γιατί αυτό βέβαια το πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στην απρόσκοπτη ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πλην όμως, πλην εάν η μη θέση εφαρμογή ή η κακή μεταφορά σε εθνικό δίκαιο ε, των οδηγιών μπορεί μερικές φορές να πηγάζει από κακή πρόθεση του κράτους μέλους, ε, ενδέχεται και να προκύπτει από προβλήματα συνοχής ή σαφήνειας του νομοθετικού κειμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν πάντοτε να ε, καταδικάζουμε για τα προβλήματα αυτά μόνο τα κράτη-μέλη. Ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι πλήρης βέβαια πληροφοριών, πλην όμως δεν επιτρέπει να εντοπιστούν ακριβώς τα προβλήματα στις ε, ελλείψεις, τα ελλείμματα μεταφοράς. Και γι' αυτό πέραν των αριθμητικών δεδομένων πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει μια ποιοτική προσέγγιση και να εντοπίσει περισσότερο τους λόγους για τους οποίους τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται ως προς τη θέση εφαρμογή της μίας της άλλης οδηγίας. Ω εκ τούτου, πίνακα αποτελεσμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει και μέσον άσκηση πίεση προ τα κράτη-μέλη, αλλά και ένα εργαλείο που θα επέτρεπε καλύτερα να ε, ερμηνεύουμε τα προβλήματα, τι δυσκολίε, ε, τι ιδιαίτερε συνθήκε που έχουν τα κράτη-μέλη. Με κάποιου δείκτε ενδεχομένω θα μπορούσαμε να δίνουμε περισσότερε πληροφορίε και για τι ε, προθεσμίε, για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, αλλά και τι ιδιαίτερε δυσκολίε τη καθοδηγία. Και όπω λέει και η θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε κινδύνους ε, για ελληματική ε, μεταφορά σε εθνικό δίκαιο μια οδηγία. Έτσι λοιπόν, μαζί με τα κράτη-μέλη, θα πρέπει η Επιτροπή να βοηθά σε όλη τη διαδικασία τη θέση εφαρμογή, έτσι ώστε να αποκλείονται δεχόμενα προβλήματα και ή, αν εμφανίζονται να επιλύονται πριν από την εκπνοή μια προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Έτσι λοιπόν, κάποιο ο οποίο θα έχει το κύρος και τι ικανότητε να παρέμβει στην ε, ε, διαδικασία αυτή τη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητο να διοριστεί σε επίπεδο των οργάνων μα, ε, όπω λέει ο κύριος Κόκ όπως άλλωστε έχει προβλέψει μια τροπολογία του στην έκθεση. Και επίση ο κύριος Κόκ λέει ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συνοχή μεταξύ του πίνακα αποτελεσμάτων τη ιστορική αγορά και του σχετικού που αφορά την αγορά σε επίπεδο καταναλωτού. Όπω άλλωστε αναφέρει και η συγγήτρια στην έκτη παράγραφο. Πιστεύει όμω ο κύριος Βανκόκ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περισσότερο συντονισμό των εργασιών στου δύο αυτού τομεί στα γερμανικά τώρα. Αυτό είναι το κείμενο το οποίο μου έδωσε ο συνάδελφος και πιστεύω ότι ε, αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτά τα οποία είπε και η κυρία εισηγήτρια. Πολύ σημαντικό δηλαδή είναι στο πλαίσιο αυτό να ε, συντονιστούν καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, τα νομοθετήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εσείς αναφερθήκατε και στο Solvit, αλλά γενικά πρέπει να έχουμε καλύτερο συντονισμό για πιο αποτελεσματική δουλειά. Είναι μια πολύ καλή θετική προσέγγιση η δική σας, πιστεύω. Οι δε πίνακε αποτελεσμάτων θα μπορούσαν, ε, αρχικά βέβαια έχουν ε, ε, προβλεφθεί για να εντοπιστούν τα προβλήματα, αλλά μπορούν σε μια δεύτερη φάση να αποτελέσουν και παράγοντα αποτροπής των προβλημάτων και εν τέλει επίλυσης και ε, βελτίωσης των αποτελεσμάτων μας. Το επόμενο ε, βήμα λοιπόν θα ήταν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο, να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι πίνακες αποτελεσμάτων και αυτό βέβαια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δυνατόν και καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε Εύελιν. Ευχαριστώ για αυτή την τόσο ε, ευφυή ανάλυση του θέματος. Πάντως μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι κάτι που σαφώς απασχολεί και την Επιτροπή μας. Θα φροντίσουμε να το τονίσουμε αυτό και στον κύριο Μόντι. Το θέμα των ποιοτικών ε, στοιχείων, της ποιότητας, είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε και σε σχέση με την αμοιβή αναγνώριση των προσόντων. Όλες οι χώρες προσπαθούν να μεταφέρουν αυτή την οδηγία που υπονοεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ποιότητα του αρχικού κειμένου. Όλοι λοιπόν κοιτάζουμε τι σχετικά προβλήματα υπάρχουν και ίσω είναι και ένα από του δείκτε που θα χρειαστεί να συμπεριλάβουμε στο μέλλον. Κύριο Ρίπεγκαρτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τούν για το εξαιρετικό της έργο και την πολύ ωραία αυτή έκθεση. Ήταν πολύ ευχάριστη η συνεργασία μαζί σας. Και πρέπει να πω ότι συνολικά την έκθεση τη στηρίζουμε. Ωστόσο θα ήθελα να αποβάλω κάποιες τροπολογίες και θα ήθελα να συνεχίσω στα δανεικά, εάν μου επιτρέπετε. Βάλτε λοιπόν τα ακουστικά σας, παρακαλώ. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση αυτή, διότι σε καιρού κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Υπάρχουν νόμοι λοιπόν που προβλέπουν το πώ θα λειτουργήσει η εσωτερική αγορά και υπάρχουν και συνεχώ περισσότερε σχέσει, διευρωπαϊκέ, εμπορικέ σχέσει μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα μας υπό το φως αυτό. Εδώ υποζητούμε βελτιώσεις, αλλά όπως υπόθηκε, εννέα είναι οι χώρες που ξεπερνούν το όριο του 1%, του 1% και πρέπει να επιδιώξουν περαιτέρω βελτίωση. Υπάρχουν τρεις προπολογίες που θα ήθελα να σας ε, επισημάνω. Το πρώτο που μπορεί να συμβεί είναι να έχουμε... Αυτό μάλλον πρέπει να γίνει κατά πρώτον, είναι να επικεντρωθούμε περισσότερο σε συγκεκριμένους στόχους και να τους δώσουμε και κάποια προβολή. Αν θέλουμε να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους κάποιες χώρες, θα πρέπει να τις πιέσουμε σαν κακούς μαθητές να κάνουν τα μαθήματά τους. Ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε μια διαδικασία κατονομασίας, και να τις κατονομάζουμε τις χώρες αυτές προκειμένου να τις φέρνουμε στο σωστό δρόμο. Και θα μπορούσαμε να έχουμε και μια μέθοδο που να είναι και πιο φιλική προ τα μέσα μαζική ενημέρωση στην παρουσίασή τη και όχι στεγνέ στατιστικέ όπω τώρα. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον ε, δημοσίευση των πινάκων. Θα πρέπει να μπορεί και η κοινή γνώμη να τα δει αυτά με απόλυτη διαφάνεια και θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις δεξιότητες και ικανότητες των διοικητικών υπηρεσιών, των εθνικών δικήσεων. Οι διοικητέ σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι και σε θέση για να, αντιμετωπί... να φέρουν εις πέρα στην ε, μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών. Νομίζω ότι η ανταλλαγή μεταξύ των Ευρωπαίων ε, ηθινόντων θα είναι πολύ χρήσιμη. Η κυρία Τούν επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά ίσως είναι το κατάλληλο σημείο που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ίσως αυτό θα είναι μια καλή ιδέα. Επίσης νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει σε επίπεδο διυπουργικό. Και κάτι άλλο που μπορεί να γίνει είναι να θεσπίσουμε μια ομάδα υλοποίηση σε μορφή clusters ίσως ειδικών ομάδων αναχώρα που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. Με την συνδρομή αυτών των clusters ίσως να εμπλέξουμε χώρες με παρόμοια προβλήματα χωρίς να δημιουργήσουμε μία μεγάλη ε, ετερογενή ομάδα, ετερόκλητη ομάδα χωρών με διαφορετικά προβλήματα που ο καθένα θα προσπαθεί να λύσει τα δικά του από τη δική του πλευρά. Όχι, να δημιουργήσουμε κλάστες χωρών με ομοιόμορφα προβλήματα ώστε να αναζητήσουν και κοινέ λύσεις. η υλοποίηση λόγω χάρη τη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών θα μπορούσε να έρθει ει πέρα σε μεγαλύτερο τρόπο κατά αυτόν τον τρόπο. Πρόσφατα να πω ότι η οδηγία Solvit έδωσε την αφορμή στην Επιτροπή να επισκεφθεί τη Στοκχόλμη για να δει πω πάνε τα πράγματα με την οδηγία αυτή και συζήτησε με υπαλλήλου και το θέμα των ε, κονδυλίων που αφορούν την οδηγία. Στη Δανία, αν πάρω το δικό μα παράδειγμα, υπάρχει ένα γραφείο υπεύθυνο για την υλοποίηση τη οδηγία αυτή, αλλά κανεί δεν ξέρει ακριβώ τι γίνεται με του πόρου, με τα κονδύλια που πηγαίνουν και. Τέλο πάντων, με το Solvit το θέμα δεν είναι μόνο τα κονδύλια. Είναι ότι το συμφέρον των χωρών προστατεύεται και διασφαλίζεται και ότι έχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν. Ε, επίσης έγραψα μια επιστολή προς τις δανέζικες εταιρείε όπου τις προσκάλεσα να κάνουν το ίδιο. Μιλήσαμε για το ίντερνετ μόλις προλίγου και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εδώ όλα τα μέσα που διαθέτουμε ώστε να προωθήσουμε καταλήλως στην κοινή γνώμη το Solvit. Νομίζω ότι ο φυσικός εντοπισμός των γραφείων Σόλβιτ είναι ήδη κάτι που μπορεί να μα απασχολήσει. Τώρα το να βρίσκεται χωμένο σε κάποιο υπουργείο ή σε ένα back office ε, το, η αρμόδια υπηρεσία είναι δύσκολο, καθιστά δύσκολο το να μπορούν να έχουν πρόσβαση εύκολα οι πολίτες, οι άνθρωποι, ενδιαφερόμενοι οι ενώσει βιομηχανιών στι διάφορε χώρε, η δανέζικη βιομηχανία, η ολλανδική βιομηχανία. Σίγουρα θα ήθελε να έχει εύκολη πρόσφαση. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια απλή λύση και αρκετά αποτελεσματική. Τέλο για τα επαγγελματικά προσόντα, θα θέλαμε να έχουμε αποτελέσματα εγκεκριμένα Ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε ένα νέο δίκτυ για να μπορέσουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ μέγιστης εναρμόνισης και ελάχιστης εναρμόνισης από την άλλη. Αυτό θα μας ε, επιτρέψει να εντοπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί δεν καταφέρνουμε να έχουμε βέβαια αναγνώριση των επαγγελματικών προσώπων, προσόντων ως τώρα. Ίσως έτσι να φωτίσουμε καλύτερα και τους λόγους, τις πηγές των προβλημάτων. τι υποκρύπτουν αυτές οι δυσκολίες στο μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε ίσως ε, πιο αξιόπιστες πληροφορίες για το όλο θέμα και αυτό να μας ε, διευκολύνει. Με αυτά τα σχόλια ήθελα να επιβεβαιώσω για μια φορά την πρόθεσή μου να συνεργαστώ στενά με την εισηγήτρια και του υπόλοιπου εισηγητέ. Ευχαριστώ. Έχω τον κύριο Ρούλε τώρα και για να κλείσουμε με του ε, και μετά ο κύριο Φαπ και ο κύριο. Κύριε Ρούλε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μας ε, για την έκθεση. Είναι καλή ιδέα, ιδιαίτερα αυτή η πρόταση για το Φόρουμ της Εσωτερικής Αγοράς, τη συνεργασία δηλαδή με τους διάφορους φορείς και παράγοντες που εμπλέκονται στην υπόθεση τη ε, ε, της μεταφοράς των οδηγιών. Τα όσα είπαν εκεί προαναλύσαντες είναι πολύ χρήσιμα. Θα ήθελα σε ένα σημείο μόνο να επισημάνω που και ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αν μιλούμε για μεταφορά σε εθνικό δίκαιο, ουσιαστικά μιλούμε και για νομοθεσία. Η νομοθεσία έχει πάντοτε ε, διαφορετική ποιότητα τα νομοθετικά κείμενα. Άρα ίσως χρειαστεί και να διατυπώσουμε επικρίσεις ε, ως προς τα νομοθετικά κείμενα και γι' αυτό ε, ίσως θα πρέπει να παρακολουθούμε την τους λόγους για τους οποίους δεν έχει γίνει η ορθή μεταφορά σε ε, εθνικό δίκαιο των οδηγιών. Ίσως θα ήταν σκόπιμο αντί να κοιτάμε συλλήβδιν ε, το θέμα της ε, μη έγκαιρης ή της μη ορθής εφαρμογής, να ρίχνουμε μια πιο συγκεκριμένη ματιά στους λόγους για τους οποίους δεν έχει γίνει η εφαρμογή αυτή, όπως την περιμέναμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούλε. Ασφαλώς το θέμα των λόγων της κακής εφαρμογής έχουμε πολύ δουλειά ακόμα να κάνουμε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ο κύριος Μπίλαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και εσάς που είχατε την ιδέα. της πρόβλεψης μιας συνάντησης ε, με τον κύριο Μόντι, ο οποίος έχει μακρά εμπειρία και πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα αυτά να διαδραματίσει. Θα είναι πολύ ε, χρήσιμη λοιπόν αυτή η συνάντηση. Και μια και ε, εκφράζω σε ευχαριστήσεις. Με ευχαριστώ και την κυρία Τσούν ε, πάνω απ' όλα για την διάθεση συνεργασίας που επέδειξε καθώς βλέπουμε ότι η έκθεση αυτή έτυχε τέτοιου τύπου συνεργατικής επεξεργασίας που θα μπορούσε να αποτελέσει και πρότυπο για τους άλλους συγητές. Για δε την δημοσίευση του πίνακα των ε, αποτελεσμάτων για την ιστορική αγορά, ε, συμφωνώ μαζί σας ότι όντως έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή της κρίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξεταστεί, τα συμφραζόμενα αν θέλετε, έχουν μεγάλη σημασία. Η δημοσίευση του πίνακα, ναι, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Οι στόχοι που έχουν προσδιορίσει από το 2006 οι κυβερνήσεις δηλαδή το ε, μέγιστο έλλειμμα μεταφοράς του 1% είναι στόχος που πρέπει να επιδιώκουμε βέβαια, που πρέπει να επιτευχθεί βέβαια, αλλά ξέρουμε ότι ακόμη 9 είναι οι χώρες που δεν έχουν επιτύχει τα ποσοστά αυτά. Ε, και μεταξύ αυτών των 9, 9 δυστυχώς εγκαταλέγεται και η Πολωνία που εκπροσωπώ εγώ. Ε, τούτου λεχθέντος Έχουμε και μεγάλο πρόβλημα ως προς την, ε, τον κατακαιρματισμό της ε, νομοθεσίας, διότι δεν ε, γίνεται ομοιόμορφα η εφαρμογή μιας οδηγίας στο επίπεδο του ευρωπαϊκού δικαίου. Και πολύ σωστά προτείνει η συγγήτρια δύο πίνακες αποτελεσμάτων, δηλαδή έναν για την εσωτερική αγορά και έναν για, την, για τον καταναλωτή, να τους δημοσιεύουμε ταυτόχρονα έτσι ώστε να οργανωθεί σωστά και το φόρουμ για την οστερική αγορά. Αυτή η πολύ καλή πρωτοβουλία της, της ε, εισηγήτριας, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα φόρουμ συζήτησης, ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, αλλά και ένα φόρουμ μέσα από το οποίο θα ασκηθούν πιέσει στα κράτη-μέλη, ειδικά αυτά τα οποία δυσκολεύονται προς την θέση εφαρμογή κάποιων οδηγιών. Πιστεύω επίση ότι θα πρέπει να ξεκολουθήσουμε να πιέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να απαιτήσουμε πιο λεπτομερεί ε, πληροφορίε ω προ ε, τα προβλήματα στη συμμόρφωση των κρατών μελών. Από τα τελευταία μας συνεδρίαση θυμάμαι ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είχε πει ότι το έγγραφο που έχει στη θέση της Επιτροπή είναι μόνο εσωτερικό έγγραφο. Συμφωνώ όμως με την εισηγήτρια ότι οι εν λόγω πληροφορίες ε, θα πρέπει και να διατίθενται ανοιχτά, δημόσια, για τον κάθε πολίτη, ώστε να είναι σε θέση να ενημερώνεται, αλλά και να είναι πιο λεπτομερής. Και ίσως είναι καλή λύση το, ε, η ιστοσελίδα ε, που θα επιτρέπει τη λεπτομερή ενημέρωση. Ωστόσο, πέραν αυτή τη πολύ καλή λύση, υπάρχει και μια άλλη λύση πολύ καλή, την οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει επαρκώ, το Solvit δηλαδή. Εμεί πάντα λέμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη χρηματοδότηση, αλλά και καλύτερη οργάνωση του Solvit. Γιατί υπάρχουν περιοχές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση στον πολίτη. Ο πολίτης δεν έχει δει πουθενά το Solvit. Δεν έχει διαφημιστεί, δεν έλεγα αρκετά το Solvit. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριος Βάπ και κύριος Μπαρνία μου στο λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Με κάλυψαν οι προαλήσαντες αλλά θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά, για την ε, ετήσια αυτή έκθεση. Ε, βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε και νέες ιδέες και φρέσκες ιδέες και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Σημειώνω ότι οι πίνακες αυτοί μπορούν να αποτελέσουν μία μόνο απεικόνηση της πραγματικότητας της εφαρμογής της εσωτερικής αγοράς και να βοηθήσουν ε, τα κράτη-μέλη στην βελτίωση των επιδόσεών τους. Πριν όμως είναι περίπλοκη η εικόνα ως προς την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και γι' αυτό είναι και δύσκολο να την αντιληφθούμε στο σύνολό της. Αυτά τα οποία προτείνει και η κυρία Τούτ με το, με το συσχετισμό με το φόρουμ για την εφαρμογή της εσωτερική αγοράς είναι μια πολύ καλή πρόταση ασφαλώς. και δίνει εν μέρη και ε, απάντηση προς το ζήτημα των ε, παραβάσεων της, ε, παραβιάσεων μάλλον της, των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και, το, ε, και θα μας επιτρέψει να δούμε πόσο περίπλοκη είναι για τον καταναλωτή αλλά πάνω απ' όλα για την επιχείρηση και για, τον, για, για, για τις αρχές της δημόσιας η εφαρμογή ε, μερικές φορές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για τον επιχειρηματία λοιπόν, για τον καταναλωτή, πάνω απ' όλα πρέπει να μεριμνήσουμε να έχουμε μια ορθά λειτουργούσα, μια ε, ε, εύχρηστη θα έλεγα νομοθεσία, πράγματα τα οποία βεβαίω εμείς ως πολιτική ομάδα πάντοτε υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπαρνί έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. χωρίς να θέλω να γρηγορήσω, ε, θεωρώ ότι όλο αυτό το πίστη της αμυναπολικής πλευράς πάρα πάρα πολύ σημαντικά και μπράβο για το έργο που επιτελέστε. Έχουμε εδώ πέρα τώρα την αντιπαράθεση ε, όλων των, των ενδιαφέρον πλευρών, των ε, εμπορευμένων, των καταναλωτών και από πλευράς εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει να σας πω ότι ε, ακριβώς ε, υπάρχουν δυσκολίες που ανεφέρθηκαν από τους προορίσαντες. Εμείς προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την επίδοσή μας για την ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών, αλλά όπως ξέρετε κινούμεθα στην μετριότητα, γιατί πολλές φορές έχουμε ε, καθυστερήσεις, έχουμε οδηγίες που φτάνουν, φτάνουν την ώρα που υπάρχει φόρτος κοινωνικής εργασίας. Άρα το κλειδί όσον αφορά την την αποτελεσματικότητα είναι το να υπάρχει συνεργασία ε, μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου. Η, η νομίζω ότι τα διερεύνησε όλα πάρα πολύ καλά, τις δυνατότητες που μας προσφέρει της Λισαβόνας και έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει τέτοιου είδους προσέγγιση. Άρα θα πρέπει. Ε, δεν λέω να γίνεται αυτό κάθε τρεις και λίγο, αλλά να βρισκόμαστε με την Εθνική Κοινοβούλια. Και έτσι κάθε τον τρόπο να υπάρχει μια τέτοιου είδου ε, ε, διαίρεση των αρμοδιοτήτων και της κυριαρχίας του ΣΥΠΗΝ μεταξύ του ενός κοινοβουλίου και του άλλου. Άλλωστε, άλλωστε όταν 15-20 χώρε έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με μια οδηγία, ε, είναι προφανέ γιατί. Είναι ένα κείμενο το οποίο αφορά τι ειδικέ επιτροπέ, αφορά τις, ε, τα εθνικά κοινοβούλια και ε, ενδεχομένω γι' αυτό το λόγο θα πρέπει μία φορά το χρόνο να βρισκόμαστε. Και δεν είναι θέμα τη αμφισβήτηση ε, είναι θέμα τη δημοσιότητας, δημοσιοποίησης, είναι θέμα κουλτούρα που θα πρέπει να, να, να μεταλαμπαδευτεί. Έτσι νομίζω ότι ο κόσμος θα μπορέσει να συμμετάσχει περισσότερο στα ευρωπαϊκά πράγματα και νομίζω ότι η κυρία Τούν θα πρέπει αυτό το δηλαδή, υπόψη όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, όλους τους συναδέλφους και ιδίως την κυρία Τούν. Πριν δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα σα πω το εξή πρώτα-πρώτα. Ε, αυτό το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά που αναφέρατε συζητήθηκε από τους συντονιστε και συζητήθηκε να υπάρχει ένα φόρουμ ενιαίας αγοράς. Αυτό ε, μου θυμίζει τότε, κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, κυρία Γκέβγαρτ, υπό την προεδρία της κυρίας ε, Παλάθιο είχε αναλάβει η κυρία Γκέπχαρτο μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα. Επομένως, σε συνέχεια της έκθεσης εκείνη ίσως θα πρέπει να ε, έρθουμε σε επαφή με τον νέο επίτροπο ή την νέα επίτροπο για να δούμε τι μπορεί να γίνει για ένα τέτοιο φόρουμ για την ενιαία αγορά. Φαντάζομαι πιο σωστό χώρο είναι αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Επίση, όσον αφορά γενικότερα ε, την εσωτερική αγορά και τη μεταφορά των ευρωπαϊκών διατάξεων στην εθνικό Ίσως θα γνωρίζετε από τις πολιτικές ομάδες ή θα το μάθετε ότι έχουμε δύο θέματα όσον αφορά την μεταφορά της αμοιβίας αναγνώρισης, της σχετικής οδηγίας, όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες και τη μεταφορά της και αυτά θα ζητηθούν τέλη Νοεμβρίου στην επομένη Ολομέλεια. Θα συζητηθούν με Συμβούλιο και Επιτροπή. Όλα αυτά βέβαια θα συζητηθούν στις πολιτικές ομάδες και ελπίζω να συμμετάσχετε εσείς όλοι εκεί ζωηρά. Επομένως, το Κομισιόν έχει το λόγο και κατόπιν θα δευτερολογήσει, θα κλείσει συζήτηση κυρία Τούν, Κομισιόν. Ενρικ Νέρκ λέγομαι. Ασχολούμαι με την εσωτερική αγορά. Εγώ και η παρακαθήμενη συνάδελφος. Έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας. Όσο αυτό βρίσκονται συμφωνώ με τα όσα άκουσα, νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε με την εισηγήτρια. Ε, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε, να δούμε τι είδους ε, καινοτομίες μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το scoreboard. Έχουμε και αυτό το ετήσιο φόρουμ, καλή ιδέα. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε το Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτό το νέο φόρουμ ε, να γίνεται σε ετήσια βάση και συμφωνώ με όσους ανέφεραν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας ε, ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μια αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των προτέρων. Να μην τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα δηλαδή και να αρχίζει η αντιδικία με τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, χρειάζεται να γίνεται ορθά και να γίνεται και έγκυρα. Και στη συνέχεια ε, να επιβάλλεται, να εφαρμόζεται επιτόπου αυτό το κοινοτικό κεκτημένο. Είναι πάρα πολύ βασικό επίσης. Όποτε έχουμε κάποιες προκλήσεις, όλα διακυβεύονται στο επίπεδο της μεταφοράς του εθνικού δικαίου στα κράτη-μέλη. Και βέβαια πάρα πολύ βασικό είναι η τήρηση από τους πολίτες. Βεβαίως και υπάρχουν διαφορές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Άλλο θέμα είναι η ποιότητα της νομοθεσίας. Ε, βεβαίως το πρέπει να βάλει την υπόψη πολυπλοκότητας της πραγματικότητας. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας παραπέμψω σε μια σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά κάποια εταιρική σχέση με τα κράτη-μέλη. Αυτό έγινε πρόσφατα και κατά τη γνώμη μας σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, σε εταιρική σχέση με τα κράτη-μέλη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ε, επιχειρήσεων και των πολιτών. Και αυτό να γίνεται εκεί, επί Άρα να δούμε τι γίνεται στα κατημέρια, τι γίνεται με τις κρατικές υπηρεσίες που πρέπει να εφαρμόσουν το κοινωτικό δίκαιο στην πράξη. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και βέβαια, αν εσείς βοηθήσετε, θα είναι καλοδεχόμενη κάθε σας βοήθεια. Το Solvit είναι ένα μηχανισμό επίλυση προβλημάτων, όπω θα ξέρετε, που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Και έχουμε σήμερα χίλιε υποθέσει ετησίω. Το Solvit ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Άρα έχει επιδόσεις εντυπωσιακέ. Όπω είπε κάποιο βουλευτή, είναι θύμα της επιτυχίας του. Γιατί έχουμε τόσε υποθέσει που πρέπει να φροντίσουμε. Και αυτό φέρνει δυσκολία σε σχέση με τους πόρους που έχουν στη διάθεσή μας. Και από πλευράς χρημάτων και από πλευράς ανθρωπίνων πόρων. Και από πλευράς προβολής αυτού του έργου. Και εδώ, επομένως, και σε αυτό το επίπεδο για το Solvit, κάθε σας βοήθεια καλοδεχούμενη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ λυπάμαι που δεν σα παρουσίασα νωρίτερα, αλλά στη σημειώση μου δεν αναφερόταν το ότι είστε εδώ. Ευχαριστώ που ασχολείστε. Κυρία Τούν, θέλετε τώρα να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις. Πάρα πολύ επικοδομητικές. Για μένα νομίζω είναι πάρα πολύ θετική εμπειρία να εργάζομαι εδώ, να συνεργάζομαι με τους δυο και μου φαίνεται πάρα πολύ συναρπαστικό το τι μας περιμένει στο μέλλον. Έχουμε αυτό το φόρουμ. Έχουμε την στενότερη συνεργασία. Ε, πρέπει να έχουμε πιο, ε, πιο καλό σκόρμπορτ όπου θα φανούν τα καλύτερα αποτελέσματα. Και το καλό όλα αυτά της εσωτερικής αγοράς. Εμεί ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Για να δούμε τώρα το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά το έργο σα. Σε με πληροφορίε που έχω, έχουμε την ε, καταληκτική ημερομηνία για τροπολογία στην επομένη Τρίτη ή στις 12 το μεσημέρι. Αυτό νομίζω ότι ισχύει, και είναι σωστό. Άρα, επίση θα ξανασυζητήσουμε και θα ψηφίσουμε 1η Δεκεμβρίου. Ίσως βέβαια αλλάξει αυτή η ημερομηνία ανάλογα με τις ακροάσεις που θα ακολουθήσουν, να δούμε τι θα γίνει και με την εκθέση 11 11 του μεσημέρι, πάντως αυτό να θυμάστε. Συναδελφοί είναι η ημερομηνία, προθεσμοί για τις τροπολογίες. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα συναδελφοί και έχουμε μείνει λίγο πίσω. Τώρα έχουμε δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με την εισηγήτρια την εισηγήτρια κυρία Ρούλε όσον αφορά την έκθεσή της. Αν δούμε τι διαδικασία προβλέπετε, τι θέλουμε να κάνουμε για αυτή την έκθεση. Ποιοι είναι εδώ από τους και ηγητέ. Έγκελ. Α, να, να, σε βλέπω. Παρίσταστε για το ΕΛΚ. Κυρία Γκέμπχαρτ. Κρόιτσμαν και εγώ. Αν μου επιτρέπετε θα λάβω το λόγο για λογαριασμό της εποχής μου ομάδας και ο κύριος Σαββίνη επίσης είναι εδώ και όποιος άλλος θέλει το λόγο βεβαίως και μπορεί να το πράξει. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ρίλε. Έχουμε επίσης και τον κύριο Βίτνερ που είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Κυρία Ρίλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και χαίρομαι που είμαστε παρόντες όλοι οι σκιώδεις. Ε, μέχρι, μέχρι τώρα μόνο διμερός τους είχα δει τους σκιώδες. Αλλά τώρα νομίζω μπορούμε να συναντηθούμε και να προετοιμάσουμε την ακρόαση που βλέπετε για τον Ιανουάριο. Πρόκειται να γίνει η ακρόαση λοιπόν μέσα στην Επιτροπή μας με το θέμα αυτό και με στόχο να προβλέψουμε ως οριστική προθεσμία τον Απρίλιο ή Μάιο για την υποβολή της έκθεσής μου στην Ολομέλεια. Τώρα πια που ευτυχώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία κυρίω τη ε, συνθήκης Λισαβόνας θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ, πολύ προσεκτικά τις ε, συνέπειες της εφαρμογή και βέβαια για το κοινό ιδιαίτερη σημασία έχει και το self-government εν προκειμένου, η αυτοδιοίκηση των ε, κοινοτήτων. Self-government στα αγγλικά γιατί είναι δύσκολη η μετάφραση του όρου στις λοιπές ε, γλώσσες. Έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο την αυτοδιοίκηση και πιστεύουμε ότι θα πρέπει μαζί με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ε, εμπλακούν ουσιαστικά στην υπόθεση αυτή και ε, παράλληλα να ενισχυθεί η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Αναφέρομαι λοιπόν και στην νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από το 2007 έχει προσδιορίσει, έχει διευκρινίσει κάποιους τομείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φερρυπίν στην έκθεση Μακάρθι, στη Βάιλερ έχουμε και εμείς ήδη ε, επισημάνει κάποιες ασάφειες στο δίκαιο που εντωμεταξύ έχει η νομολογία του δικαστηρίου αλλά και ε, η νομολογία του δικαστηρίου διευκρινίσει στην ε, υπόθεση Μπραμπάντου παραδείγματι στην υπόθεση του Αμβούργου. Έτσι λοιπόν αναφέρεται ότι μπορούν και από κοινού οι κοινότητες να ασκούν το δικαίωμα τους, αλλά ταυτόχρονα και ατομικά μπορούν να συμμετέχουν σε μια κοινή ομάδα συνεργασίας, σε μια κοινή δομή συνεργασίας. Υπάρχει λοιπόν διευκρίνηση του τομέα αυτού, υπάρχει επίσης διευκρίνηση του τομέα της σύμπραξης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, όπου και πάλι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είπε και η κυρία Βάιλερ νωρίτερα, έχει διευκρινίσει ότι ε, δεν χρειάζονται διπλές φάσεις τους ε, στις προκηρύξεις και επίσης υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κριτήριο της ανάληψης κινδύνου, θέματα που θα δούμε και με την ακρόαση, θέματα που έχουν να κάνουν και με τα ύδατα και με την Ιταλία, την και γενικά τις εκχωρήσεις. Ε, που δεν καλύπτονται πάντα από την οδηγία περί ε, δημόσιων διαγωνισμών, αλλά με τα, που πρέπει να συμμορφούνται, εν πάση περιπτώσει, με τα κριτήρια της εσωτερική αγοράς. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα και ο κατάλογος των ζητημάτων που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Στο ενδοτικό ή ήπιο λεγόμενο δίκαιο έχουμε αρκετά ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε επισημάνει ότι υπάρχει έλλειμμα, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, ως προς τα κοινωνικά κριτήρια και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε ένα εγχειρίδιο για το θέμα αυτό. Υπάρχει επίσης το Fair Procurement, ε, μια δημοσίευση της Επιτροπής για την ε, ισότιμη προς, ε, πρόσβαση στους δημοσιογονισμούς, αλλά και η ιδέα του Green Procurement, δηλαδή η οικολογική διάσταση στους, στις δημόσιες προμήθειες όπου θα πρέπει βεβαίως και για τις ε, κοινότητε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει ε, η βεβαιότητα ότι ε, μπορούν να δράσουν αυτόνομα και στο ενδοτικό δίκαιο. Με την έννοια του ενδοτικού δικαίου ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφύγουμε την εντύπωση ότι ενδοτικό δίκαιο σημαίνει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Όχι. Άρα θέλουμε καλύτερο συντονισμό, θέλουμε περισσότερη ασφάλεια δικαίου, αλλά και συντονισμό σε επίπεδο επιτροπής για τον τομέα των ε, προμηθειών. Και πιστεύω ότι και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγοράς έχει ρόλο να διαδραματίσει προ την ε, ασφάλεια δικαίου. Έχω υπόψη μου ε, ε, σε ένα άλλο τομέα ε, κοινότητες οι οποίες χρειάζεται να, για να εξασφαλίσουν, να τηρήσουν μάλλον όλους τους όρους των δημοσίων διαγωνισμών ως προς κάποια ε, νομική πραγματογνωμοσύνη να δαπανίσουν το 1 τρίτο του σχετικού προπολογισμού του και επιπλέον έχουν σημαντική εσωτερική επιβάρυνση και γραφειοκρατικό φόρτο, πράγματα τα οποία θα του επιτρέπουν να λειτουργήσουν όπω θα ήθελαν. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε. Θα πρέπει να δούμε και το πρόβλημα του κατακαιρματισμού τη αγορά που θέλουμε να αποφύγουμε ασφαλώ. Θέλουμε να προαγάγουμε την καινοτομία και τι νέε φάνταστε λύσει και θα ήταν καλό με τα labels, στην ε, ε, σήμανση που θα μπορούσαμε να συστήσουμε ειδικότερα με την Επιτροπή, να δούμε τι είδους κριτήρια εναρμόνισης θα μπορούσε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να είναι πιο σαφή τα κριτήρια μέσω της σήμανσης, ώστε και ο ενδιαφερόμενος ε, να γνωρίζει ποιοι κανόνες ισχύουν, να έχει την ασφάλεια δικαίου και να γνωρίζει με ποιον συνελάσσεται ή τι πρέπει να υποβάλει αυτά, ώστε να έχουμε περισσότερη ασφάλεια δικαίου, σαφήνεια δικαίου στους, ε, ε, στις προκηρύξεις. Και ίσως θα μπορούσαμε και να καταγράψουμε τις συνθήκες που ισχύουν τώρα στον τομέα αυτών να μια απογραφή αν θέλετε, ένα απολογισμό της κατάστασης. Και ένα άλλο σημείο για να κλείσω, είδαμε με την ε, κρίση ότι μπορούμε χάρη στις δημόσιες προμήθειες και τους διαγωνισμούς να δώσουμε σημαντική όθηση στην οικονομία μας. Αλλά αυτό με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφάλεια και κανόνες σαφείς για όλους. Ευχαριστώ και εγώ ίδιος και άλλοι θα έχουμε να κάνουμε παρατηρήσεις εδώ, πράγμα που δείχνει και τη σημασία του, της έκθεσης αυτής. Ο κύριος Έγγελ πρώτα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μου διότι έστω και με κάποια βραδύτητα μπορέσαμε σε στενές να οργανώσουμε μεταξύ σκιωδών εισηγητών μια επικοινωνία με την εισηγήτρια. Και μετά από τις ε, παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Ρούιλε, βλέπουμε ότι η έκθεσή της ήδη περιέχει θεμελιώδη συστατικά, κατά την εκτίμησή μου, ιδίω το στοιχείο της ασφάλειας δικαίου διότι εδώ είτε μιλάμε για οικονομικούς είτε για, δημόσι... για οικονομικούς παράγοντες είτε για δημόσιες αρχές αυτό είναι μια από τις βασικές αιτίε διαφωνίας προς στιγμή. Αυτή τη στιγμή θα φαινόταν παράξενο να μην περάσουμε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες και απλώς να διευθετήσουμε το θέμα του εφαρμοστέου και της υλοποίησης. Αυτό αφορά πολλούς τομείς και έχει άμεση σχέση και με, τον, με την έννοια του soft law, του ενδοτικού δικαίου. Είναι λοιπόν σημαντικό εδώ να ξεχωρίσουμε τις συνετές συμβουλές και τις άλλες έννοιες από τις καλές πρακτικές, το τι μπορεί να γίνει στην πράξη και ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνει και αυτή μια κατάσταση σύγχυσης όπου κανείς δεν θα καταλαβαίνει τις έννοιες για τις οποίες μιλάμε εδώ. Υπάρχουν πρακτικές που έχουν παγιωθεί πλέον και κάποια ορολογία ιδίως τους διαγωνισμούς με οικολογικό περιεχόμενο βλέπουμε να επηρεάζεται η απόφαση των δημόσιων αρχών. Ε, Εφόσον ε, λοιπόν επιδιώκουν ε, συμβάσεις, χρησιμοποιείται διαφορετική ορολογία από τις δημόσιες αρχές χωρίς να ξέρει ούτε ο ένας το άλλο για ποιο πράγμα μιλάμε και τελικά εγκρίνεται μια σύμβαση οικολογικού περιεχομένου με πολλές ελλείψει. Euh, euh, ο τομέας λοιπόν της ασφάλειας δικαίου είναι πρωταρχική σημασίας για την ε, τωρινή μας πορεία και επεξεργασία της έκθεσης. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να δούμε τα οικολογικά στοιχεία με τρόπο προσεκτικό προκειμένου να φροντίσουμε και την πρόοδο της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτή την κατεύθυνση. Μια άλλη μέρημνα που συχνά μας απασχολεί, ιδίω ε, λόγω της παρουσίας των εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δεν φαίνεται να διαφωνούν με την ενίσχυση της οικολογικής διάστασης που θα ήθελαν όμως να μπορούν να έχουν και πλήρη συμμετοχή βάσει κανόνων ξεκάθαρων και που να ισχύουν με τρόπο ισότιμο για όλους. Πέραν αυτών, για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα ήθελα να σταθώ εδώ, να σταματήσω εδώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που θα μπορέσω στο άμεσο μέλλον να έχω τόσο στενές συναντήσεις με την εισηγητρία. Ε, Κύριε Κεπχαρτ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Μπερνιό, η οποία επίσης ε, λόγω της απεργίας δεν μπορούσε να είναι εδώ. Αλλά δεν μπορώ εγώ, μια καλή σοσιαλδημοκράτησα, να διαμαρτύρομαι για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας από τον εργαζόμενο, θεωρώ τόσο σημαντική, σημαντικό. Και έτσι θα αντικαταστήσω την κυρία Μπερνιό ε, χωρίς ε, Πριν όμω περάσω στο γαλλικό κείμενο που μου έδωσε στην συνάδελφο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Ρούλε για τι προσπάθειέ τη και για τι επιλογέ τη, γιατί βλέπω ότι έχει επισημάνει κάποια πάρα πολύ σημαντικά σημεία, πολύ θετικά σημεία. Έχει δώσει δηλαδή ήδη μια κατεύθυνση για την ακρόαση, την οποία, τα οποία θεωρεί ευπρόσδεκτα ιδιαίτερα η δική μου η ομάδα και στα οποία φυσικά θα συμπράξει το βαθμό του δυνατού. Θα ήθελα ξεκινώντα να πω ότι θα πρέπει πάντα να κινούμεθα πλέον από εδώ και μπορώ ε, στο πλαίσιο της ε, συνθήκη της Λισαβόνας και να καταγράφουμε τα ε, επιτεύγματά μας. Βεβαίως της, την πρόοδο προς το θέμα της λειτουργίας των πρωτοβάθμιων τοπικών αρχών, της αυτοδιοίκησης και να υπογραμμίσουμε, όπως άλλως το πράξετε και εσείς, την, ε, τα, τα, νέα εργαλεία που μας προσφέρει η συνθήκη για την ε, λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν τα οποία είναι τόσο σημαντικά. Και θα πρέπει ασφαλώς ε, να τα δούμε τα έγγραφα αυτά, τα θέματα αυτά στις διαστάσεις τους σωστές. Μιλήσατε εσείς ήδη για το ενδοτικό δίκαιο για τις διάφορες ανακοινώσεις και τις διάφορες προσεγγίσεις που έχουν κατά καιρούς εκφραστεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύω ότι θα πρέπει εν τέλει στα συμπεράσματά μας να απευθύνουμε μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τακτοποιήσει τα διάφορα θέματα σε σεβασμό βέβαια των συνθήκων που ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει όλα αυτά πλέον δηλαδή να μπουν σε μια σειρά μαζί σας, με την συγκήτρια δηλαδή, ε, ξέρω ότι αυτό το έγγραφο, αυτή η δουλειά βρίσκεται σε καλά χέρια και θα προχωρήσει αποτελεσματικά. Τώρα μου επιτρέπετε θα περάσω στα γαλλικά και πάλι για να κάνω ανάγνωση του κειμένου του συναδέλφου. Ε, χαίρομαι που μπόρεσα να συνεργαστώ στην έκθεση του πρωτοβουλίας με την κυρία Ρούλε την εισηγήτρια, ε, με την οποία πιστεύω ότι έχουμε ο τέλος συμπληρωνόμαστε στις θέσεις μας. Η εισηγήτρια μας ξέρω ότι είναι στρατευμένη σε θέματα κοινωνικά και κριτήρια περιβαλλοντικά στο πλαίσιο των ε, δημοσίων προμηθειών. Ε, πρόκειται πράγματι για θέματα κέρια σημασία, τα οποία και εγώ εδώ τεράστια ε, σημασία και θα ήθελα πέραν αυτό να συμπληρώσω και κάποια άλλα σημεία στην έκθεση. Θεωρώ δε ότι η κυρία Ρούλε και οι συνάδελφοι θα ήταν καλό να εξετάσουν τα ζητήματα αυτά. Θεωρώ λοιπόν πρωταρχικής σημασίας το να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες και ε, ιδιαιτερότητες των τοπικών ε, και περιφερειακών αρχών και των εδαφικών μονάδων των διαφορών εδαφών στην ε, επικράτεια των κρατών μελών. Επίσης, και για να απηχούμε και τις συζητήσεις ε, που έλαβαν χώρα χθες το πρωί, πρέπει να προσδιοριστούν ιδιαίτερε ε, διαδικασίες και προθεσμίες ως προς την καταβολή των ποσών ε, στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές οι καθυστερήσεις για την καταβολή των αντιτίμων από πλευράς των τοπικών αρχών μπορεί να έχουν πολύ σημαντικό, σημαντικές επιπτώσεις για τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν πρέπει βέβαια αυτό να σημαίνει και σημαντική επιβάρυνση των τοπικών αρχών. όπω άλλωστε υπογράψαμε και χθε. Και τελευταία παρατήρηση που θα θέλω να διατυπώσω για να ληφθεί υπόψη είναι για μένα ιδιαίτερα σημαντική και έχει να κάνει με τη λήψη υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των κοινωνικών, των υπηρεσιών ε, κοινή ωφελία. Δεν μπορεί δηλαδή η ανάθεση, η δημόσια ανάθεση να υπακούει μόνο στι έννοιε τη ιδιωτική αγορά και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Γιατί πρέπει να εξασφαλιστούν, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν ποιοτικέ καθολικέ υπηρεσίε στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών και όχι μόνο με καθαρά λογιστικού όρου. Αυτά είναι διάφορα σημεία στα οποία ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε εντελεχέστερα κατά την επεξεργασία της εκθέσεως και ευχαριστώ τους συναδέλφους και την συγκήτρια για την προσοχή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γεφαρδίου Πρόεδρος. Τώρα για την άλλη, ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καταρχάς χαίρομαι που ασχολείται με το θέμα αυτό η κυρία Ρούλε είχε ήδη πει και στο παρελθόν ότι οι δημόσιες αναθέσεις και μέσα από την νομοθεσία αλλά και πάνω απ' όλα μέσα από την ομολογία παίρνουν τώρα μια διαφορετική μορφή και πρέπει να συστηθούν ε, διεξοδικά. Τώρα πιστεύουμε ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε και την έμφαση και του στόχου τη συζήτηση. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ισότιμε συνθήκε ανταγωνισμού για τι επιχειρήσει, τι δημόσιε προμήθειε, ε, κατά την προκήρυξη των διαγωνισμών από τι δημόσιε υπηρεσίε. Πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο ευνοϊκέ συνθήκε ε, ε, σε επίπεδο στο δυνατόν πιο κοντινό στις κοινότητες με, με τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση σε γραφειοκρατικό φόρτο και θα συστήσουμε φυσικά με την ε, εισηγητρία ενδεχομένω και, το και το ενδεχόμενο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ηλεκτρονική μορφή της επικοινωνίας και της ε, διεξαγωγής των ε, διαδικασιών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες κοινότητες που έχουν μείνει πίσω σχετικά με την ηλεκτρονική αυτή δυνατότητα. Άλλες οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο Αλλά υπάρχουν πολλοί δήμοι και κοινότητε που δεν αξιοποιούν ακόμη τις δυνατότητες προσφέρει το ε, ηλεκτρονικό σύστημα. Όμως θα έπρεπε πιστεύω να προχωρήσουμε με περισσότερη έμφαση σε αυτή τη διάσταση διότι εξοικονομούμε και χρόνο αλλά και χρήμα. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι όταν είναι μεγάλο ο γραφειοκρατικό φόρτο, η επιβάρυνση οικονομική για μια επιχείρηση η οποία αναλαμβάνει λόγω τη ε, ε, μη ικανοποιητική γραφειοκρατική οργάνωση επεδοκινότητα ε, έναν ε, διαγωνισμό, ήδη αυτή η επιχείρηση μετά θα μεταφέρει την, το κόστο αυτό στον καταναλωτή ασφαλώ. Γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Και τώρα να σας μιλήσω εγώ ως και ηγητής. Πρόκειται για ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό τμήμα του έργου της Επιτροπής μας, κυρία Ρουλέ. Χαίρομαι που τον ελάβατε γιατί μπορείτε να τα καταφέρετε σε αυτό το θέμα. Πρέπει όλοι να εργαστούμε και να βοηθήσουμε τώρα των συντονιστών γιατί θα ασχοληθούμε αυτό το θέμα την επόμενη πενταετία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα πρώτα-πρώτα. Ε, αναφέρεται την έκθεση της κυρίας Βάιλερ και άλλες εκθέσεις. Αλλά πρέπει να θυμηθείτε και την έκθεση Harbor για τις ε, συμβάσεις προανταγωνισμού. Οπότε μην το ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε αυτό που είχα γράψει εκεί, γιατί όταν θέλουμε θέσει απασχόληση θέλουμε και καινοτομία, ε, πρόκειται για κάποιους πόρους που έχουν μια εκμετάλλευση. Άρα στις εκθέσει ε, θυμηθείτε αυτά τα οποία είχα προτείνει, δανειστείτε ιδέες και όπως είπε ο κύριο Έγκελ, ο κύριο Κρότσμαν, και άλλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υπόθεση αυτή. Αυτό το πρόβλημα ταλαιπωρεί πολλά κράτη-μέλη. Υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας σε πολλές χώρες. Και στη δική μου χώρα. Πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία. Και θέλουμε να εμπλακούν στην κοινοτομία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι άλλο που δεν αναφέρθηκε όμω ήταν το πώς θα γίνει η μεταφορά τη οδηγία για τα ένδικα μέσα. Αυτό έχει ήδη συζητηθεί και ήταν τμήμα της προσπάθειας του να πείσουμε τις εταιρείε ότι προχωράμε όπως πρέπει. Η διαδικασία προχωρεί και ότι τις φροντίζουμε κατά κάποιο τρόπο. Κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει με την Σουηδία. Πήγαμε εκεί, συναντήσαμε τις αρχές της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό και μας είπαν οι αρμόδιοι ότι ασχολούνται και με τις ε, δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες. Και θεώρησαν ότι αυτό είναι στην και εκ των ονού για να είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και αγορά τους. Άρα ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι κάνει το κράτος και οι κρατικές αρχές πάνω σε αυτό. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ φιλόδοξο, αλλά ας είναι το πλαίσιο της ε, δουλειάς μας στο μέλλον. Θα ξαναλάβει το λόγο κυρία Ρίλα, δούμε και το χρονοδιάγραμμα. Αυτά είχα να πω εγώ και ο και ο κύριος Σουβάμπ έχει το λόγο, αλλά και η κυρία Βάιλερ. Και κατόπιν ο κύριος Βίτνερ από την Ορμόδια Γενική Διεύθυνση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τόσα υπόθηκαν. Κύριε Ρούλη, Ρούλη πράγματι έχει ε, κάνει μια πολύ καλή επισκόπηση των θεμάτων που, πρόκειται να, που πρέπει να συζητηθούν Όντως έχουμε νέα δεδομένα από τη συνθήκη της Λισαβόνας και για τις ε, τοπικές αρχές. Θα επικεντρωθώ εγώ στα λίγα που με ενδιαφέρουν περισσότερο, γιατί τα λοιπά έχουν καλυφθεί. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ασφαλώς ε, θα πρέπει να συζητηθεί και ιδιαίτερα η υπόθεση του Αμβούργου. Εδώ έχει οδηγήσει αυτή η νομολογία σε συγκεκριμενοποίηση των δεδομένων, πράγμα το οποίο θεωρώ θετικό, αλλά και σε ε, περισσότερη ασφάλεια για τις ε, κοινότητες, γιατί μπορούν να προβλέψουν τι και σε ποιο βαθμό μπορούν να κάνουν ε, στο μέλλον. Ωστόσο, υπήρξε Ε, αμφισβήτηση του κατά πόσον το περιεχόμενο της ίδιας της νομολογίας αυτής, της υπόθεσης, της απόφασης αυτής, ε, είναι σύμφωνο με την ιστορική αγορά και θα θέλαμε να το επαληθεύσουμε. Επίσης, ως προς το κατά πόσον μπορεί η κοινοτική αρχή να στηριχθεί σε κάποιους όρους που ορίζονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν είναι πολύ σαφές αυτό, δεν είναι πολύ απλή η ε, διαδικασία αυτή και το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη να καταβάλει, όπως είπε η κυρία Ρούλε, η τοπική αρχή μερικές φορές και το 30% του ε, προϋπολογισμού της ε, για να εξασφαλίσει την νομική πραγματογνωμοσύνη ως προς την ε, προσαρμογή ή την τήρηση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου αποδεικνύει πάνω απ' όλα ότι δεν υπάρχει η τεχνογνωσία δεν είναι ανεπτυγμένη ακόμα η τεχνογνωσία. Ίσως ε, στο μέλλον με περισσότερη ανάπτυξη της διάστασης ευρωπαϊκής και χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, να έχουμε λιγότερο δαπάνες για τέτοιου είδους ζητήματα. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να δοθεί έμφαση και στους ε, κοινωνικούς στόχους, στόχους κοινωνικής πολιτικής, που εξυπηρετεί μια δημόσια προκήρυξη και θα πρέπει επί τη ευκαιρία της και για τη σχετική με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να δούμε ποιοι είναι οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να διατυπώνονται αυτές ε, οι προκήρυξεις επί παραδείγματι ελάχιστες ε, προδιαγραφές ως προς τον μισθό, ελάχιστος μισθός. Ε, αν και διαρωτώ εάν είναι δυνατόν δυνάμε τις νομολογίες του δικαστηρίου να θεωρήσει ε, μια επιχείρηση προερχόμενη από άλλο κράτος μέλος ότι μπορεί να ε, παραβιάσει την αρχή του ελάχιστου μισθού ε, και παρόλα αυτά να παραμένει σύμφωνη, σύνομη με, την ευρωπαϊκή αγορά, με την εσωτερική αγορά. Πάντω είναι πολύ καλή ιδέα για την έκθεση και ελπίζουμε μέσα στον επόμενο, στις αρχές του επόμενου έτους ε, να μπορέσουμε και να την εγκρίνουμε. Ευχαριστώ κύριε Βάιλερ. Κύριε Ρούιλε, θα φαντάζεστε ασφαλώς ότι θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η προσέγγισή σας και η πρόταση του ταχύτερο δυνατό να γίνει η συζήτηση για την έκθεση, όπως άλλωστε είπα κύριε Κέπχαρτ, έχετε από πλευρά μα λάβει και το πράσινο φως σε τελευταία ανάλυση για τις προτάσεις που έχετε υποβάλει. Θα ήθελα λίγο να προτείνω κάποιες λεπτομέρειες, εν μέρη με κάλυψε ο κύριος Σφάπ. Θα ήθελα καταρχάς λοιπόν να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες προξενούν μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο η επιβάρυνση στις τοπικές αρχές λόγω της υπαρξής τους. Ίσως είναι αυτό ε, ένα φαινόμενο που καταγράφεται σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι πάντοτε και παντού. Ίσως κάπου οι νεότεροι υπάλληλοι μιας ε, υπηρεσίας κάποιου δήμου κοινότητα κοινότητας να είναι λιγότερο ενημερωμένοι, ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλους τους δήμους και κοινότητες. Επίσης, θεωρώ ότι και σε εθνικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο, και στην Γερμανία και στην Ιταλία, το βλέπουμε άλλωστε και στη Γαλλία, είναι λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ε, άκαμπτες ε, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Χοχτήφ, για, το, για την έκθεση της κολονίας. Θέματα δηλαδή τα οποία ε, βλέπουμε να κρίνει με πολύ απόλυτο τρόπο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ θα έπρεπε να περιμένουμε την εξέλιξη τους, την μεταξέλιξή τους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι τα εθνικά κοινοβούλια και οι ειδικοί στα κοινοβούλια που, ή στο κοινοβούλιο που ασχολούνται με το δίκαιο των δημόσιων προμηθειών και των προκηρύξεων θα μπορούσαν και δεν θα αναφέρουμε μόνο στη Γερμανία γιατί ίσως θα μπορούσε κάποιο άλλο κράτος να εμπλακεί να εξετάσουν ειδικά τις, ε, αυτού του τύπου τις δυσκολίες. Λυσμονήσαμε πέραν του κύριου Χάρμπορ και τον συμπαθητικό εκείνο Γάλλο συνάδελφο που είχε κάνει την οδηγία, την έκθεση για τις οδηγίες. ναι, ναι, τον κύριο Φρουτό, πολύ σημαντικό θεμέλιο της εργασίας μας εδώ. Και επίσης μιλήσατε κυρία Ρούλε και για τις οικονομικές και τις κοινωνικές τις οικολογικές διαστάσεις, αλλά εγώ θα ήθελα να δω και τα λοιπά κριτήρια. Και ναι, μπορεί να μιλούμε για τα κοινωνικά και οικολογικά όσα σημαντικότερα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τα υπόλοιπα κριτήρια. Ίσως θα έπρεπε να δούμε... το πώς προχωρεί ο διάλογος για τον ανταγωνισμό ο ανοιχτό διάλογο. Είδαμε στο Ανόβερο παραδείγμα ότι υπάρχουν κάποιε προσπάθειες, ένα μεγάλο φόρουμ, θέματα τα οποία μας ε, ανοίγουν νέου δρόμου ενδεχομένω για συζήτηση και για λύσει. Και πέραν αυτού του μεγάλου ανοιχτού διαλόγου θέλουμε να Ε, ανοίξει το ζήτημα της λήψης των αποφάσεων έτσι ώστε να μην λαμβάνει μια, ε, ένα μικρό διευθυντήριο, ένα περιορισμένο διευθυντήριο της αποφάσεις και ο λαός να μην είναι καν ενήμερος. Τα θέματα όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να τα δούμε παράλληλα και σε σύγκριση και με τη χρηματοπιστική κρίση. Θα ήταν χρήσιμο να δούμε εάν μπορούμε να ε, διδαχθούμε και να προχωρήσουμε για το μέλλον. Ξέρω ότι είναι πολλές οι παρατηρήσεις, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν όλες στην εκθέσή σας. Αλλά ίσως θα ήταν καλό με την ευκαιρία να τις συζητήσουμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε κύριε Βάιλερ. Ευχαριστούμε και για την όλη σας εργασία για αυτό το θέμα. Πολλοί είναι ενδιαφερόμενοι. Είναι σίγουρα θα σας είναι ευχάριστο να συνεργαστείτε. Ο κύριος Βίντνερ τώρα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σας παρακαλέσω να είσαστε αρκετά σύντομος, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στο μέλλον. Και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Ρούλε, για να μπορέσει να ανακεφαλαιώσει. Γιατί η κυρία Κλάση και η κυρία Σαρτόρη θέλουν να ξεκινήσουν και με το δικό του θέμα. Κυρία Βίντλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι όντω πολύ σύντομο. Η έκθεση επικεντρώνεται σε δύο βασικά ζητήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή που εξέλιξε. Η συνοχή πρώτα απ' όλα και η σχέση δημοσίων προμηθειών με άλλες πολιτικές, όπως του περιβάλλοντος, η κοινωνική και της καινοτομία. Είναι σημαντικά ζητήματα αυτά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚΤ και άλλες γενικές διευθύνσεις ασχολούνται με αυτά τα θέματα και θα ήθελαν να, υπήρξε, να υπήρχε ένα έγγραφο καθοδήγησης ενδεχομένως, ώστε όλα αυτά να παρουσιαστούν παράλληλα και να φανεί ότι τα λαμβάνουμε υπόψη και δίνουμε μια συνολική καθοδήγηση για όλα αυτά τα περίπλοκα και αλληλένδετα ζητήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές ιδέες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Επίσης η νομολογία που πολύ γρήγορα δημοσιεύεται και αναπτύσσεται για την συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιο τομέα κυρίω. Η νομολογία είναι αντικείμενο ανάλυσης και σκοπεύουμε να την αναλύσουμε, να την εξετάσουμε περαιτέρω για να δώσουμε περισσότερη γνώση και στις συμβαλόμενες αρχές. Θα συνεργαστούμε λοιπόν όσο μπορούμε περισσότερο μαζί σας από την πλευρά της Κομισιόν για να έχουμε μια ολοκληρωμένη έκθεση. Σας ευχαριστούμε πραγματικά και εμείς ανεπομονούμε για τη συνεργασία μας. Κυρία Ρούλε, έχετε κάποια καταληκτικά σχόλια. Πολύ σύντομα. Επισημαίνω πρώτα απ' όλα στους ε, σκιώδεις ότι έχω σημειώσει τέσσερις σελίδες παρατηρήσεις από τα όσα άκουσα. Προφανώς και θα τα ε, διηθήσω και θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά. Ε, πρώτο από όλα βέβαια και σημαντικό βήμα είναι η ακρόαση. Ως προς την ε, οδηγία για την ε, αποζημίωση, η Remedies Directive, δεν αναφέρθηκα σε αυτήν γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δεν έχει, για τα ένδικα μέσα. Δεν έχει ε, λήξει ακόμη η προθεσμία για τη θέση εφαρμογή και γι' αυτό μπορώ να κάνω μία μόνο περιστασιακή ε, παραπομπή, αλλά δεν μπορώ να αναφερθώ διεξοδικά στην οδική αυτή. Πάντως φυσικά προσβλέπω στην ε, ακρόαση την οποία θα οργανώσουμε από κοινού με τους συναδέλφους και τους συγκητές και, τον Ιανουάριο, για τον Ιανουάριο και βέβαια και τις τροπολογίες σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλη σας την συμβολή και να επιβεβαιώσω ότι το χρονοδιάγραμμά μας προς στιγμή είναι ακρόαση είτε στις 25-26 Ιανουαρίου θα ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες ώστε το δυνατόν συντομότερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους γι' αυτό και περνάμε στο τελευταίο μας σημείο για αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, θέση στην εμπορία μάλλον και χρήση των βιοκτώνων προϊόντων. Με ιδιαίτερη χαρά μου καλωσορίζω την κυρία Κλάς, εισηγήτρια του θέματος αυτό από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, σας καλωσορίζουμε θερμά και τη δική μας εισηγήτρια την κυρία Σαρτόρη, η οποία ηγείται των εργασιών μας για την ετοιμασία της νομοδότησης αυτής. Μια πολύ ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των δύο επιτροπών. Σήμερα ένα βασικό ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι ότι ζητήσαμε από την Επιτροπή ανακεφαλαίωση της μελέτης αντικτύπου για το θέμα αυτό. Θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι αυτό έχει γίνει παγιωμένη τακτική στην Επιτροπή μας. Η κυρία Σαρτόρη μάλιστα ζήτησε να γίνει αυτό και για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε θα έλεγα να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή ευθύ αμέσω να παρουσιάσει το, τη μελέτη αντικτύπου και μετά να δώσω το λόγο στι εισηγήτριες και να κάνουμε τη συζήτησή μα. Νομίζω ο κύριος τον Μπορέτσι, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σα, που είναι επικεφαλή υπηρεσία στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο και υπεύθυνο για το θέμα αυτό, θα παρουσιάσει την ε, μελέτη αντικτύπου του φακέλου σα, Κανονικά έχετε μια ανακεφαλαίωση όλη των μελέτη αντικτύπου. Πέντε σελίδε, όμω, το σύνολο, οι 80 σελίδε τη μελέτη αντικτύπου, μπορούν να διατεθούν από τη γραμματεία σε όσου το επιθυμούν. Στα αγγλικά όμω. Ξέρω ότι οι συγκίτρε γνωρίζουν πολύ καλά το έγγραφο, αλλά αν χρειαστεί να δούμε τα δεδομένα, να έχουμε υπόψη ότι είναι στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σχεδόν, σχεδόν σωστά το είπατε. Ευχαριστώ τέλο πάντων που σα απασχόλησε το θέμα. Πρέπει να ευχαριστώ και την κυρία Σαρτόρη, διότι επέδειξε αυτό το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτή τη γνωμοδότηση, διότι η πρόταση είναι πολύ σημαντική. Επίση, με μεγάλη μου χαρά, ε, βλέπω ότι ασχολείται με αυτό και η κυρία Κλάς. Οπότε για να κάνουμε ε, να ρίξουμε μια ματιά ε, στο τι γίνεται εδώ και τι γίνεται με τη μελέτη των επιπτώσεων. Πρώτα πρώτα δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι θέλουμε να έχουμε μια οδηγία άλλη που, που, που ακολουθεί την προϋπάρχουσα επί μια οκταετία. Έχει γίνει εν μέρη ικανοποιητική, εν μέρη ορθή εφαρμογή της, αλλά εν μέρη ήταν αναποτελεσματική, ήταν ελληματική εφαρμογή της και το, το θέμα ήταν να πετύχουμε στόχους για την υγεία, για το περιβάλλον, για κάποιες ε, ουσίες που θα έπρεπε να άποσουν από την αγορά και τώρα γνωρίζουμε καλύτερα τι γίνεται με τα βιοκτώνα, τι γίνεται με, με, με, με τι άλλες ουσίες υπάρχουν στην αγορά, κάτι το οποίο δεν ίσχυε προηγουμένως και αλλά υπήρχαν και κάποια κρατημέλη τα οποία δεν είχαν καθόλου νομοθεσία όσον αφορά τα προϊόντα τα σχετικά με τα βι-οκτώνα Και έτσι κυκλοφορούν στην αγορά. Οπότε αυτή η οδηγία η οποία ισχύει εδώ και μία οκταετία είχε κάποιο θετικό αποτελεσμα. Όμως ταυτόχρονα, ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι η τιμή, το τίμημα ήταν υψηλό. ηταν αναποτελεσματικό της, ήταν κάποιες τιμές ιδιαίτερα υψηλές γιατί οι εταιρείε που ασκούσαν την εμπορία, οι εταιρείε που έκαναν την παραγωγή ήταν αυτοί που ονομάζονται formulators, τέτοιου είδου. Κάποιο είδου τέλο πάντων ΜΜΕ και είχαν την αρχική ουσία την οποία παρήγαγαν ε, κάποιε, σε μερικέ περιπτώσει, μεγαλύτερε εταιρείε που ήθελαν να μπορέσουν να καλύψουν το υψηλό κόστο. Και θα έπρεπε να γίνει πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον, η υγεία και να ενισχυθεί η βιομηχανία τόσο ώστε να θέτουν σε εμπορία προϊόντα με αποτελεσματικό τρόπο. Όπως προαναφέραμε, έχουμε εδώ πέρα δύο βασικούς στόχους. Πρώτα-πρώτα το να μειώσουμε το κόστος συμμόρφωσης που ήταν πολύ υψηλό και έχουμε την απουσία υποχρεωτικής κοινοποίησης δεδομένων και επίσης θέλαμε να βελτιώσουμε το περιβάλλοντος και υγείας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια παραθυράκια στην ισχύουσα οδηγία, τα οποία παραθυράκια θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν. Και ένα εντυπωσιακό παράδειγμα είναι κάτι το οποίο έχει γνωρίσει η δημοσιότητα εδώ και κάνα χρόνο. Ότι δηλαδή, όταν έχουμε ένα καταναλωτικό προϊόν, το οποίο σχετίζεται, έχει δηλαδή στοιχεία βιοκτώνου, μπορεί κανείς να το θέσει σε εμπορία μόνο αν υπάρχει έγκριση αυτή τη βιοκτονουσία. Όμως, εάν αυτό το καταναλωτικό προϊόν εισάγεται στην Ευρώπη, δεν προβλεπόταν, δεν υπήρχε ενίσχυε καμία διάταξη ελέγχου τούτου του προϊόντος. Καναπέδες και παπούτσια ήταν βασικά προϊόντα σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Είχαν σχετιστεί κάποια από αυτά τα προϊόντα, τα εμπορεύματα, με ουσίες που ήταν τέτοιες που είχαν προκαλέσει εγκάβματα. Χιλιάδες καταναλωτών πήγαν στο νοσοκομείο σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Να, ένα παράδειγμα του πώς θέλουμε να ενεργήσουμε προς προστασία της υγείας με το νέο νομοθέτημα. Της υγείας και του περιβάλλοντος τώρα και ένας άλλος στόχος ήταν το να συρρυκνώσουμε τις δαπάνες και το κόστος. Βέβαια, έχουμε αυτή τη μελέτη των επιπτώσεων που καλύπτει διάφορα, διάφορες πηγές και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι πετύχαμε τη συρρυκνώση της δαπάνης και του κόστους, εκτός από αυτά τα, τα, τα, τα προϊόντα που έχουν περάσει από χημική επεξεργασία. Έχουμε και την ετικετοθεσία αυτών των ε, κρατονικών προϊόντων που να λέει δηλαδή η ετικέτα ότι έχουν υποστεί επεξεργασία με βιοκτώνα. Τώρα υπάρχει αυτό ως προαπαιτούμενο, ως, ως, ως προοδοτική ρύθμιση, κάτι το οποίο δεν ίσχυε προηγουμένως. Οπότε, αυτό τώρα ειδοποιεί, προειδοποιεί και αυτούς που έχουν αλλεργίες. Στα παπούτσια δε δεν ήταν ε, θέμα καν του αν είσαι αλλεργικός. Όποιος φόραγε εκείνα τα παπούτσια ε, υφίστατο σωματική βλάβη. Αύξηση μόνο τη δαπάνη γινόταν και πετύχαμε την συρρήκνωσή της. Α, έχουμε και άλλο παράδειγμα. Θέλουμε δηλαδή να είναι πιο ενδελεχής η διαδικασία της αδειοδότησης για το προϊόν. Σαφέστερη, σαφέστερη διαδικασία. Να, παράδειγμα. Όσον αφορά τι προθεσμίε, τώρα είναι πιο πιεστικέ. Δεν υπήρχε προηγουμένω προθεσμία τόσο ώστε να εγκρίνει κάποιο κράτο μέλο το τελικό προϊόν. Τώρα υπάρχουν δεσμευτικέ, πιεστικέ προθεσμίε. δεν είχε ιδέα η κάθε εταιρεία, η κάθε επιχείρηση πότε θα εγκριθεί το προϊόν της. Αυτό δεν ήταν καλό βέβαια. Δεν μπορούσαν να κάνουν προγραμματισμό οι εταιρείε και οι βιομηχανίε. Ούτε αυτοί που κάνανε την έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα, ούτε αυτοί ξέρανε τι, τι, τι, τι νομικό, τι χρονικό συγγνώμη, πλαίσιο ισχύει. Αυτό το παράδειγμα και άλλα πολλά θα μπορούσε να βρει κανεί αν ήθελε. Επίση, προβλεπόταν ένα σύστημα το οποίο αποσκοπήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τόσο είναι πιο κατευθυνό, κέντρο κατευθυνόμενη η έγκριση και υπάρχουν τα παράλληλα συστήματα κατά κάποιο τρόπο, διότι παράλληλα μπορούν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να χορηγούν τι εγκρίσει, όπω σα ε, οδήγησα, σα εξήγησα και με, με, με σαφέστερε, με πιεστικότερε προθεσμίε, αλλά υπάρχει η διαδικασία, υπάρχει η πρόληψη για κάποια προϊόντα να πάνε σε αυτή την πιο κεντρική διαδικασία, δηλαδή να περάσουν τα προϊόντα από την υπηρεσία του Ελσίνκη. Μιλούμε για χημικά προϊόντα. Μιλούμε για αποτελεσματικότητα κλίμακας που πετυχαίνεται έτσι και έτσι θεωρούμε ότι θα επιταχυνθεί η κατάσταση, η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο εξωθούμε τις μικρότερες επιχειρήσεις να κινηθούν προς καινοτομία. Επίσης, θέλουμε να καλύψουμε όλα τα προϊόντα τα οποία σχετίζονται με τις νέες ουσίες, όποιες μπουν στο παιχνίδι, στην αγορά, στο μέλλον. Ένα άλλο στοιχείο, πολύ σημαντικό. Επιτρέπουμε ακόμα στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τη διαδικασία έγκριση σε εθνικό επίπεδο. Οπότε, από την άλλη μεριά, ενισχύθηκε η αμοιβαία αναγνώριση. Ούτω ώστε να διαφωνηθούν εταιρείε στην αγορά. Επομένω, αν κάποιο κράτο μέλο δώσει το πράσινο φω για κάποιο προϊόν με βιοκτώνα, τότε τα άλλα κρατημέλια είναι υποχρεωμένα να εγκρίνουν το ίδιο προϊόν, εκτό εάν μπορούν να αιτιολογήσουν την άρνησή του. Εδώ υπάρχει συγκρισιμότητα με την νομοθεσία για τα ε, παρασιτοκτόνα. Και τα ζυζανιοκτόνα. Μιλούμε για κάποια αγορά με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. προϊόντα για, για, την επιμελητία στα καράβια μέχρι εντομοκτόνα ε, προϊόντα που σχετίζονται με τη γεωργία, ε, ζυζανιοκτώνα για πάρκα των πόλεων κλπ. Μιλάμε για τεράστια ε, τεράστια εύρος προϊόντων, αλλά κυρίως μιλάμε για κάποιο είδους βιομηχανικά προϊόντα, όπου ε, ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση από ό,τι τα ζυζανιοκτώνα. Οπότε και γι' αυτό φροντίσαμε αυτή την νομοθεσία. Και αυτό το αναγνώρισε η μελέτη των επιπτώσεων. Επίσης, υποχρεωτική, υποχρεωτικό, υποχρεωτική κοινοποίηση δεδομένων σε σχέση με κάποια ζωικά προϊόντα. Αλλού χρειάζεται επίκληση παλαιότερων δεδομένων, αλλού όχι. Και είπαμε να έχουμε τέτοια προσέγγιση τόσο ώστε να είναι κάπως τα πράγματα λιγότερο γραφειοκρατικά και έτσι να μπορούν οι εταιρείε και τα προϊόντα να κινηθούν ευκολότερα, να είναι πιο εύκολο το σύστημα. Και ξέρετε, μέσα αυτήν την οχταετία μόνο ένα-δύο προϊόντα εγκρίθηκαν στην δυνάμει αυτού του συστήματο. Και επίση έχουμε προτείνει μια εναρμονισμένη δομή για τα τέλη σε εθνικό δίκαιο, μια δομή, δηλαδή όχι σε ένα επίπεδο, αλλά σε μια δομή, να κατανέμεται, να κατανέμονται τα τέλη. Ταυτόχρονα θα πρέπει, όπως και με το ΡΙΤΣ, να ε, προσδιορίσουμε μέσω της επιτροπολογίας την νομοθεσία της σχετική με τα τέλη και προτείνουμε ε, μείωση τελών για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. μετατρέπουμε το κείμενο από οδηγία σε κανονισμό και για να αποφύγουμε την ε, καθυστέρηση από μια μεταβατική περίοδο, αλλά και για να περιορίσουμε το γραφειοκρατικό φόρτο και επίσης, το πιο σημαντικό, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη τήρηση τόσο των διατάξεων όσο και των προθεσμιών. Διατάξεων που θεωρούμε σημαντικέ και για τους ορισμούς και για τις προθεσμίες, για να μπορούν οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις να δράσουν σε μια διευρυμένη και ε, εύρυθμη εσωτερική αγορά. Ε, σταματώ τώρα γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μακρηγόρησα και ευχαριστώ να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Σας ευχαριστούμε. Ήταν ε, πολύ χρήσιμη η συνολική αυτή παρουσίαση μιας τόσο σφαιρικής προσέγγισης. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι η περίληψη μας παρουσιάσατε Σίγουρα δεν μπορεί να εκθέσει όλη την αξία τη μελέτη αντικτύπου και αυτό συμβαίνει συχνά με τι περιλήψει. Υπάρχουν σημεία του κειμένου τα οποία θα πρέπει να ε, τονιστούν σωστά με έντονου χαρακτήρε λόγω χάρη να φανούν οι επιλογέ που κάνατε στην περίπτωση που υπήρχαν πάνω από μία. Στη σελίδα 48 λόγου χάρη, εάν δείτε το κείμενο της μελέτης αντικτύπου, αναφέρεται ο τρόπος ανάλυσης του κόστους Θα ήταν πολύ καλό λοιπόν να ξέρει κανείς τις λεπτομέρειες για να καταλάβει την ε, εξισορρόπηση κόστους και κινδύνων που έχετε, κόστους ωφελίας που έχετε διεξαγάγει. Πάντως είναι πάντων χρήσιμο να έχουμε έστω και μια γραπτή περίληψη των, ε, μιας τέτοιες μελέτης και όλων των ανάλογων μελετών για την Επιτροπή μας. Και μια τεχνική παρατήρηση, αυτό ήταν μια τεχνική παρατήρηση. Από την πλευρά του Προέδρου σα, ποιο θέλει τώρα πρώτα στο λόγο, η κυρία Σαρτόρη ή κυρία Κλάση. Η κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικά σχόλια προκαταρκτικά για το περιεχόμενο της μελέτης. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι όπως ακριβώς το θύμισε μόλις η εκπρόσωπος της Επιτροπής, έχουμε στα χέρια μας ένα νομικό εργαλείο, έναν κανονισμό για τέτοιους ε, σκοπούς έχει φανεί μέχρι τώρα ότι αυτό είναι το καταλληλότερο νομικό μέσο και για την άμεση εφαρμοσιμότητά του για την άμωση μάλλον εφαρμογή του σε κάθε κάτος μέλος και γιατί διορθώνει αναδρομικά και κάποια άλλα προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένας λόγος για να είμαστε ήδη ικανοποιημένοι. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα ήθελα να θυμίσω εδώ όπως ζήτησε ο κύριος Άρμπουρ με την επιστολή του της 22ης Ιουλίου του 2009 στην συνδιάσκεψη των Πρόεδρων υπάρξει μια κατάλληλη μελέτη της κατανομής των αρμοδιοτήτων σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Ζητήθηκε κάποια κεφάλαια να εξεταστούν μεμονωμένα. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακόμη με βεβαιότητα πώς, τι έκβαση είχαν οι διαπραγματεύσεις και πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή περιβάλλοντος, όμως ο συνάδελφος κλά ενδεχομένως να μας δώσει μια επιβεβαίωση. Έχουμε στενή συνεργασία για να συζητήσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά, τα αυτά σε κάθε περίπτωση. Και θα συναντηθούμε για να ορίσουμε τις λεπτομέρειες και τις κατανομής αρμοδιοτήτων. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα δούμε ακριβώς ποιο περιεχόμενο θα αναλάβει κάθε επιτροπή και αυτό που αναλογεί στη δική μας. Τώρα, για το σύστημα δύο επιπέδων, όπως το προβλέπει η Οδηγία του 98, αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να το ξαναδούμε και στο σύνολό της μάλιστα. Υπάρχουν πολλά αντιφατικά σημεία που παραμένουν όμως στην πρόταση και θεωρώ απαραίτητο κάποιες πτυχές να συζητηθούν περαιτέρω. Θεωρώ ότι η σημερινή διατύπωση του κειμένου θα πρέπει να μεταβληθεί. Θα σας παρουσιάσω τα σημεία στα οποία θεωρώ ότι χρειάζεται παρέμβαση. Πρώτον, τα κριτήρια αποκλεισμού. Θεωρώ ότι τα κριτήρια αποκλεισμού για ενεργές ουσίες, όπως διατυπώνονται στο κείμενο της πρότασης, στο άρθρο 5 απαιτούν καλύτερο ορισμό προκειμένου να επιτύχουμε τους επιδιωκόμενους στόχους. Πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες εξαιρέσεις για την ε, σωστή λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και με το χρόνο να έχουμε και ένα αυξανόμενο επίπεδο εισαγωγών που να προστατεύει την ε, υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλον. Ένα δεύτερο σημείο είναι η διαδικασία της εξουσιοδότησης, της κοινοτική στην πρόταση περιελήφθη μια κεντρική διαδικασία, κοινοτική διαδικασία για την εξουσιοδότηση, την οποία δέχομαι θετικά, διότι πρόκειται να δημιουργήσει ένα σύστημα θεωρητικά πιο ταχύ και Στι διαδικασίε αυτέ προβλέπεται ένα σύστημα διαβούλευση με τα άλλα κράτη-μέλη, το οποίο στην περίπτωση τη εθνική εξουσιοδότηση για την αμοιβαία αναγνώριση, ω τώρα έχει αποδειχθεί βραδύτερο και πιο περίπλοκο. Εάν σωστά ερμηνεύω τα κίνητρα που οδήγησαν την Επιτροπή να υποβάλει μια τέτοια πρόταση, θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλέψουμε τη δυνατότητα να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή τη διαδικασία για την κοινοτική εξουσιοδότηση και σε άλλε κατηγορίε. Σταδιακά μεν, αλλά πριν από το 2023. Αυτό το τωρινό κείμενο το αναφέρει και Προσωπικά βρίσκω ότι είναι τεράστια αυτά τα χρονικά διαστήματα, υπερβολικά μεγάλα. Επίσης το θέμα της έρευνας και καινοτομίας. Από τη μια πλευρά εμείς με αυτόν τον κανονισμό τονίζουμε ότι είναι ανάγκη να προασπιστούμε και να προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Όμως στο άρθρο 46 της πρότασης ε, ορίζεται σαφώς τι και πώς μπορεί να εκτελεχθεί σε επίπεδο πειραμάτων και επιστημονικών δοκιμών. Γνωρίζοντα το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο για όλου του τομεί που μα απασχολούν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και το τελικό κόστο των διαδικασιών. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν υπόψη ότι οι κανόνε που τώρα πάντοτε μας απασχολούν όταν μιλάμε για έρευνες, καινοτομία και δοκιμές. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι κανόνες αυτές επιβάλλουν να περικόψουμε στο δυνατόν περισσότερο το κόστος. Η τωρινή πρόταση λοιπόν θα μπορούσε να περιέχει κίνητρα για την καινοτομία και θα Πρέπει να σκεφτούμε την μεταβατική περίοδο που μπορεί να, να ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς οι επικίνδυνοι οργανισμοί θα εξελίσσονται με ταχύτητα, αναπτύσσοντας αντίσταση στα ουσίες και στα βιοκτώνα που θα χρησιμοποιούνται, αν δεν προβλέψουμε μια δυνατότητα αλλαγή των ίδιων των διαδικασιών. Τέταρτο σημείο, ανάγκη να αποσαφινιστεί καλύτερα η έννοια της διατύπωσης πλαίσιο σε σχέση με την προηγούμενη. Δεν είναι σαφές ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να περιληφθεί ένα βιοκτόνο που ανταποκρίνεται στα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά μέσα σε ένα πλαίσιο διατύπωσης που ήδη προϋπάρχει. Δεν είναι σαφέ τι θα πρέπει να έχουν υπόψη οι επιχειρήσει όταν θα αλλάξουν ενδεχομένω τα όρια ανοχή για τι ενεργέ ουσίε στο εσωτερικό μιας ήδη εξουσιοδοτημένης διατύπωσης. Εδώ χρειάζονται λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές, περαιτέρω κανόνες για να διευθυνθούν οι περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη σημερινή πρόταση. Σε ό,τι φορά την αμοιβαία αναγνώριση, είναι, καλύτερα, είναι καλύτερη η διαθέτηση που προτείνεται τώρα σε σχέση με την προηγούμενη, όμως χρειάζεται πάλι σαφέστερος ορισμός, λεπτομερέστερος και αυτό λόγω και της έλλειψης εμπειρίας που έχουμε σε σχέση με την υλοποίηση του ορισμού αυτού. Ως σήμερα, καμία διαδικασία αμοιβές αναγνώρισης δεν έχει λειτουργήσει ολοκληρωμένα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κατά πόσο χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες ώστε αυτό να μπορέσει να γίνει πράξη. Μια άλλη κατηγορία προϊόντων που απαιτούν ορισμό καταλληλότερο, προσφορότερο, είναι που, αυτοί που παρουσιάζουν τα λεγόμενα βιοκτώνα χαμηλού κινδύνου. Το άρθρο 17 εκθέτει κριτήρια τα οποία θα έπρεπε να καλύπτουν αυτού του είδου τα προϊόντα. Χρήσιμο πάντως θα ήταν κατά την απόψή μου να προσδιορίσουμε καλύτερα τις έννοιες της ε, αμεληταία έκθεσης και των, ε, των κανονικών συνθήκων χρήσης, ώστε να έχουμε ορθότερη ερμηνεία των άρθρων. Τώρα για τα υπόλοιπα άρθρα, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής είναι ένα από τα επιχειρήματα που οδήγησαν στην αναθεώρηση της οδηγίας. Εγώ είμαι, εκφράζω τη χαρά μου που μια σημαντική κατηγορία προϊόντων, όπως αυτά στα άρθρα που ανέφερα συμπεριλήφθη, για τους, στο πεδίο του προτινόμενου κανονισμού. Ιδίω το άρθρο 47, όπου εκθέτονται οι διαδικασίε επισήμανσης των ε, συγκεκριμένων προϊόντων και ισχύουν και διατάξεις που καλύπτουν άλλες κατηγορίες προϊόντων στο άρθρο 58. Συμφωνώ απολύτως με την ανάγκη ίχνη τέτοιων προϊόντων, ιδιαίτερος όταν είναι προϊόντα εισαγόμενα. Σε ό,τι αφορά την συγκριτική αξιολόγηση, για την ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων όταν έχουμε πλέον αρκετή εμπειρία για τη χρήση αυτών των νέων προϊόντων. Αυτό είναι ένα σημείο όπου ελπίζουμε ότι θα λάβουμε το μεταξύ και νέες προτάσεις. Και τελευταίο σημείο, ένα σημείο ευαίσθητο, το οποίο έχει να κάνει με την σημερινή κατάσταση του συστήματος εξουσιοδοτήσεων και το πώς λειτουργεί αυτό στην αγορά και πώς εισάγονται ενεργές ουσίες και βιοκτώνα στην αγορά. Εδώ θα έχει το χρόνο ο formulator για να δώσει την εξουσιοδότηση και να θέσει σε εμπορία ένα συγκεκριμένο προϊόν. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για εξουσιοδότηση θα μπορούν να επιλέξουν να περιμένουν την απόφαση της αρμόδιας αρχής. Οι φορείς αυτοί ονομάζονται στην αργό, την καθημερινή γλώσσα, free riders. Θα πρέπει όμως εδώ να προβλεφθούν κάποιες αλλαγές ώστε οι υπονομαζόμενοι free riders να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα όσους ε, περιμένουν τις προβλεπόμενες εξουσοδοτήσεις. Πολλοί από αυτούς είναι σαφώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται η Ευρώπη και αυτές πρέπει να υπερασπιστεί. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε ξανά τον επιδοκόμενο στόχο μας. Το έργο που μας περιμένει είναι τεράστιο, η πρόταση δεν είναι απλή και το χρονοδιογράμμα μας προβλέπει ανταλλαγή απόψεων 25 και 26 Ιανουαρίου του 2010 όταν θα έχουν ετοιμαστεί, μάλλον η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι στις 26 Φεβρουαρίου. Τώρα για το άρθρο 50 και βάσει των κανόνων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιτροπών μπορεί το χρονοδιάγραμμα αυτό να μεταβληθεί εντωμεταξύ ανάλογα και με τις εξελίξεις τις οποίες θα μας επισημάνει η συνάδελφος κυρία Κλάς. Um, Ευχαριστούμε για αυτή τη συνολική σας παρουσίαση κυρία Σαρτόρη. Θα σας αφήσουμε να επιδιώξετε εσείς τη συμφωνία για τους συγκεκριμένου τομείς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Σίγουρα, βλέποντα κανεί τη μελέτη που αντιλαμβάνεται ότι οι αλλαγέ στην εξουσιοδότηση προϊόντων και τα ζητήματα που σωστά ε, ναι, η Κομισιόν για τα εισαγόμενα προϊόντα λόγου χάρη, τα επεξεργασμένα συστατικά ή τα θέματα τη επίβλεψη αγορά, όλα αυτά απασχολούν και τέλο και την Επιτροπή μα. Τα γνωρίζουμε και μα ενδιαφέρουν και το θέμα της αμοιβέ αναγνώριση. Είμαι βέβαιο ότι όλα αυτά θα τα μελετήσετε περαιτέρω. Μπορούμε τώρα να έχουμε γενική συζήτηση και ερωτήσει προ την Κομισιόν για τη μελέτη αντικτύπου. Απλώ να βεβαιωθώ ότι οι σκιώδει συζητητέ είναι εδώ. Έχω την κυρία Γκέπχαρτ, ο σκιώδη, ο κύριο Μπεσόη δεν είναι εδώ, ο κύριο Κρόιτσμαν όμω είναι. Η ακούραστη κυρία Ρούλε, εάν θελήσετε να παρέμβετε παρακαλώ. Ο κύριος Φόξ είναι εδώ, ο κύριος Σαβίνη δεν είναι και ο κύριος Μπαρνιέ θα ήθελε να συνεισφέρει. Σύντομα σχόλια λοιπόν αν θέλετε για να έχει το χρόνο και η Επιτροπή να απαντήσει. Κυρία Κλάς, με συγχωρείτε. Σας κοιτώ, αλλά δεν είχα σκοπό να σας παραβλέψω. Θα πάρετε εσείς το λόγο αυτής αμέσως και μετά θα έχουμε τους σκιώδεις εισηγητές και τις παρεμβάσεις τους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και κύριο, ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να λάβω το λόγο στην Επιτροπή σα. Θα είμαι σύντομη, γιατί η κυρία Σαρτόρη αναφέρθηκε διεξοδικά σε όλα τα σημαντικά ζητήματα. Η αξιολόγηση του κόστου τη πρόταση αυτή από την Επιτροπή και με την κυρία Ποτσίδη μιλήσαμε και χθε στη δική μα Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Μου φαίνεται κάπω δύσκολη υπόθεση διότι διότι το θέμα αυτό δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε μόνο σε όρους ευρώ και λεπτών. Έχουμε να κάνουμε με το κέρδος ως προς το περιβάλλον, ως προς την δημόσια υγεία. Που αντίστροφα αν δεν υποστηριχθούν θα οδηγήσουν σε διαφορετική ε, κατάσταση ως προς το κόστος και τις ταπάνες. Αυτά λοιπόν. για να πω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ως προς το κείμενο στο οποίο θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν σημεία στα οποία μπορούμε να έχουμε μια καλή ε, μπορούμε να έχουμε επικάλυψη λίγο πολύ και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία για να τα αποφύγουμε και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση των επιπτώσεων, το impact assessment, ε, στο οποίο αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, και το πολύ μεγάλο εύρος, πολύ μεγάλη ψαλίδα που μας παρουσιάζει, από 193,6 εκατομμύρια μέχρι 706 εκατομμύρια, είναι ασφαλώς δύσκολο να προχωρήσουμε με κάποιον ασφαλή υπολογισμό λέει η Επιτροπή ότι αν πρόκειται να εξασφαλιστεί η εξοικονόμηση δαπανών, πρέπει αυτή να είναι πιο σωστά αιτιολογημένη. Εγώ βλέπω και από τα άρθρα που επεξεργαζόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή ενημέρωση, οτιδήποτε δηλαδή εισάγεται από τα κράτη-μέλη, από τα τρίτα κράτη να ορίζεται με βάση, να τη χάνει με βάση ε, τα όσα ισχύουν για τα κράτη-μέλη. Τώρα, εάν θα πρέπει μέσα σε κάθε προϊόν το οποίο αγοράζουμε, φερειπίν σε ένα κομμάτι ύφασμα που θα αγοράσω μέσα στην εσωτερική αγορά, να υπάρχει η σήμανση του κάθε είδους προϊόντος ή ουσίας ή ίνας που περιλαμβάνεται μέσα στο ύφασμα, αυτό δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο ή δυνατόν να το πούμε. Επίσης, παρακολουθούμε την κατάσταση του ΡΙΤ στη δική μου την Επιτροπή ως προς την εξέλιξη του, ως προς την πρόοδό του. Φυσικά επηρεάζει και αυτήν εδώ την ε, πρόταση για τα βιοκτώνα, η πρόοδος του ΡΙΤ και ίσως θα ήταν καλό να δούμε τι είδους οικονομική επιβάρυνση θα προκύψει από εκείνη την υπόθεση και σε ποιο βαθμό μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς. Η Επιτροπή τώρα προτείνει ένα σύστημα ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, χορήγηση αδειών. Πλην όμως δεν θέλω να σημειώσω ότι δεν μου φαίνεται ξεκάθαρο το ποιος ορίζει το προϊόν ε, χαμηλού κινδύνου, low risk ή high risk αντίστροφα. Πώς μπορούμε λοιπόν να περιοριστούμε μόνο σε αυτό Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να προσβλέπουμε σε καλά αποτελέσματα από τη συνεργασία μας. Τώρα έχουμε να κάνουμε μόνο ένα πρώτο βήμα και πάντω θέλουμε να έχουμε ασφαλείς προδιαγραφές και ισότιμες παντού προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν, παραδείγματι, κύριε Σαρτόρη, πάω διακοπές στην Ιταλία και αγοράσω ένα εντομοαποθητικό σπρέι, Θέλω να είμαι ήσυχη ότι το αγοράζω με, τους, με τις ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας και προστασίας της υγείας μου, όπως αυτές που ε, ξέρω ότι ισχύουν στη Γερμανία, Φερρυπίν. Αυτά και προσβλέπω, όπως είπα, στην πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Είναι πολύ καλό αυτό το εγχείρημα με πολλές ε, διακλαδώσει πιστεύω και συνέπειες προς την ιστορική αγορά. Σωστά επισημάνατε ως προς την αξιολόγηση των επιπτώσεων ότι ήταν η εξοικονόμηση πόρων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο πολύ στηριγμένη στην ε, διοικητική απλοποίηση, απλούστευση, αλλά θα πρέπει να δούμε και σε επίπεδο καταναλωτή τι είδους επιπτώσεις μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Ορισμένα θέματα σήμανσης ε, αναφέρονται μόνο σε μία μικρή παράγραφο μέσα στο κείμενο, ενώ ταυτόχρονα εμείς έχουμε ένα ευρύτερο έργο υπό επεξεργασία για τη σήμανση και ίσως ε, θα έπρεπε να το δουν διαφορετικά η κυρία Σαρτόρη και ο κύριος Μάντλς. Για να δούμε λοιπόν τώρα τους και οδησηγητές με τη σειρά και μάλιστα ξεκινώ με την κυρία Γκέπχαρτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή τη φορά είμαι η σκιώδη συγκεντρία. δεν εκπροσωπώ πλέον άλλον, παρά μόνο τον εαυτό μου. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε να κάνουμε με απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε στο σπίτι, απορριπαντικά, βιοκτώνα και άλλα. Ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων καθημερινής χρήσης. Και αναφέρονται δύο βασικοί στόχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κόστος ε, λειτουργίας του συστήματος πρέπει να είναι περιορισμένο στο βαθμό του δυνατού. Αφενός, αφετέρου δε, να είναι όσο δυνατόν υψηλότερος ο βαθμός προστασίας της δημόσιας υγείας. Για μένα, Επιτροπή, η ε, έννοια του κόστους έχει δευτερεύουσα σημασία Κύρια πρωταρχική σημασία έχει το να είμαι βέβαιη ότι όταν χρησιμοποιείτε κάποιο βιοκτόνο θα είναι ασφαλές βιοκτόνο, θα εξασφαλίζει, θα ικανοποιεί τους όρους της προστασίας του περιβάλλοντος, θα ε, είναι, ε, δεν θα ε, ρηπαίνει τον ε, υδάτινο ορίζοντα, θα είναι βιοδιαλυτό και θα είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει ζήτημα ε, προβλημάτων ως προς την ε, βιοανθεκτικότητα για να έχουμε στο δυνατόν, όπως είχαμε δει και με τα αντιβιωτικά, να μην έχουμε, ε, να έχουμε στο δυνατόν λιγότερα βιοανθεκτικά βιοκτώνα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να διευκολύνεται η εισρωή όλο και νέων βιοκτώνων από τις μεγάλες επιχειρήσεις στην αγορά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω και δεν βλέπω κανένα χείρημα που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια εξέλιξη. Επίσης θέλω να αναφερθώ ως ε, χρήσιμα μέτρα στην ε, συμπερίληψη των ε, μεταποιημένων προϊόντων, τη σήμανση, την ιχνηλασιμότητα ή ανιχνευσιμότητα, όλα αυτά τα σημεία τα οποία θεωρώ θετικά, αν και θα πρέπει να επισημάνω ότι φοβούμε, με την εμφύληξη να διαβάσω πιο προσεκτικά στο κείμενο, αν κάτι έχω καταλάβει λάθος, φοβούμε όμως ότι κάτι το οποίο ίσως ε, αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ε, light μορφή της αμοιβαίας αναγνώρισης κινδυνεύει να οδηγήσει σε περιορισμό, μείωση, υποβάθμιση των προδιαγραφών ως προς την χορήγηση άδεια για τη διάθεση στην αγορά. Δηλαδή μαζί με την αμοιβαία αναγνώριση κινδυνεύουμε να ε, μειώσουμε το επίπεδο προστασίας της δημοσιασίας και του περιβάλλοντος, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να ε, αφήσουμε να περάσει ανεξέλεγκτο. Πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Άλλωστε, πρόκειται για ζήτημα αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα όσον αφορά τη διάσταση τη προστασία των ε, καταναλωτών. Και σε αυτό συμφωνώ 100% με την κυρία Σαρτόρη. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια ε, ενισχυμένη συνεργασία και πάνω απ' όλα με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή και τη δημόσια υγεία. Και ελπίζω ότι θα έχουμε υπάρχει χρόνο μαζί με την ε, εισηγήτρια που περίμενα να με καθοδηγήσει και εκείνη για να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα αισθήματα ώστε να δεξετάσουμε τουλάχιστον τα σημαντικότερα αισθήματα επακριβώς. Και να δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα φυσικά ελάφρυνσης του γραφειοκρατικού φόρτου να την ε, υποστηρίξουμε, αλλά χωρί αυτό να θέσει σε κίνδυνο τους άλλους τομείς ε, στους οποίους αναφέρθηκα νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέπχαρτλή, ο Πρόεδρο. Κύριε Κρότσμαν, έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την Άλντε, στα αγγλικά, όπω μου ζητήθηκε θα σα πω, την γνώμη μου και κάποιε παρατηρήσει. Συμφωνούμε με το επιχείρημα της Επιτροπής δικαιολογείται έτσι θεωρήσει της οδηγίας του 98. Είναι καλά έχουμε κάθε τέτοια πρόταση που διευκολύνει τη διαδικασία. Ούτω ώστε να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και για του χρήστε και να διευκολυνθούν και οι δημόσιε αρχέ. να καλυφθούν τα προϊόντα που έχουν βιοκτώνα και να προστατευτεί έτσι η ανθρώπινη υγεία ότι για να μπορέσουμε αποτελεσματικά να έχουμε ασφαλή προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει έλεγχος των ουσιών που περιέχονται στα όσα εισάγουμε από τρίτες χώρες. Να μην επιβαλούμε έλεγχο μόνο στις κοινωτικές εταιρείε. Γιατί οι μη εταιρείε μπορούν να θέσουν στην εμπορία ότι ε, παράγουν. Μιλούμε για την ίδια αγορά και του καταναλωτέ. θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όρια ανταγωνισμού. Μην τον στρεβλώνουμε τον ανταγωνισμό. Γιατί αλλιώ οι ευρωπαϊκέ εταιρείε πηγαίνουν στι τρίτε χώρε, ώστε να μην υπάγονται σε αυτού του Τώρα, όσον αφορά την ε, διαδικασία αδειοδότηση για τα προϊόντα χαμηλού κόστου. Ε, καλή είναι και το κατευθυνόμενη διαδικασία και επίση ε, ο έλεγχο των ενεργών ουσιών. Είναι πάντως περίπλοκη η διαδικασία που υπάρχει και προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο. Μάλλον θα πρέπει να έχουμε ενιαία διαδικασία για όλα τα προϊόντα με διοκτώνα. Αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό πλευρά κόστου και πιο δίκιο για τι εταιρείε που ζητούν την ε, αδειοδότηση. Η Κομισιόν είχε πει ότι η κεντροευθυνόμενη διαδικασία θα βοηθήσει καινοτομία και έρευνα όσον αφορά τα προϊόντα αυτά. Αυτό είναι επιθυμητό. Όμως θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτή η κεντροκαθινόμενη διαδικασία να είναι απλούστερη από την ε, διαδικασία σε εθνικό επίπεδο. Η άλλως προτιθέμενη αξία δεν υπάρχει. Δεν έχει νόημα να αναθέσουμε στην ε, κοινωτική υπηρεσία που ασχολείται με τις χημικές ουσίες ε, την δουλειά αυτή, μια που έτσι απλώς θα αναλώνονται κοινωτικοί πόροι. τουλάχιστον να έχουμε ενιαία διαδικασία σε εθνικό επίπεδο. Και άρα να έχουμε ισορροπία μεταξύ πλεονεκτημάτων της κεντρικής ε, διαδικασίας και της ε, άλλης. Στα γερμανικά. κυρία Γκέπχαρτ αναφέρθηκε στον αδίρυκτο όρο, να μην ε, βλάπτεται το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Και φυσικά και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στο βαθμό του δυνατού ε, την απλούστευση τη γραφειοκρατία, αλλά εφόσον δεν υποβαθμιστεί η προστασία του περιβάλλοντο και η δημόσια υγεία. Η πρόταση Επιτροπή αναφέρει και το χαιρετίζουμε ότι στόχο τη οδηγία είναι και η βελτίωση τη προστασία της δημόσια υγεία και του περιβάλλοντο. Και άρα δεν ε, καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει όταν μιλούμε για απλούστευση, για απαλλαγή από το γραφειοκρατικό φόρτο, να θεωρούμε ότι αυτόματα αυτό συνεπάγεται υποβάθμιση τη προστασία τη δημόσια υγεία και του περιβάλλοντο. Βεβαίω, κυρία συνάδελφε, δεν μπορεί κανένα προϊόν να διατίθεται στην αγορά χωρί να έχει γίνει ε, ενδελεχή εξετασή του και βεβαίω ότι δεν είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Για μα αυτό είναι αυτονόητο. Και το υπογραμμίζουμε. Και τι θα ήταν τεράστιο σφάλμα να θεωρούμε κάτι τέτοιο, ότι δεν είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση να διατεθεί στην αγορά προϊόν το οποίο δεν είναι ελεγμένο ως ασφαλές για το περιβάλλον. Και επίσης νομίζω ότι καλό θα είναι να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η απλουστευση του γραφειοκρατικού βάρους είναι προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κάνουν την καινοτομία, που κάνουν την έρευνα, που προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις και τις οποίες πολύ συχνά λησμονούμε μέσα στην νομοθετική μας διαδικασία, ότι δηλαδή είναι εκείνες οι οποίες ακριβώς προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεν είναι δυνατόν πάντοτε να λησμονούμε ότι στόχος μας είναι και να εξασφαλίσουμε αρκετή δουλειά για τους ανθρώπους να αποδομούμε δηλαδή όλο αυτό το γραφειοκρατικό βάρος το οποίο επιτρέπει στις μικρές και μικρές επιχειρήσεις με τα καινοτόμα τους προϊόντα να προσφέρουν στην αγορά μας καθαρά προϊόντα, υγιεινά προϊόντα ε, και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν και θέσεις εργασίας για τους ε, συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά πραγματικά δεν μας μένει πολλής χρόνος. Εδώ θέλουμε να συζητήσουμε τη στρατηγική που υπονοεί η πρόταση της Επιτροπής. Το θέμα μας είναι αν είναι σωστή η στρατηγική της Επιτροπής ή όχι σήμερα. Αυτή είναι μόλις η αρχή της διαδικασίας, δεν το τέλος της. Ο, η κυρία Ρούλε. Πολύ σύντομα για να επισημάνω ότι θέτω από το προλαλήσαντα. Πιστεύω ότι σε επίπεδο ε, Επιτροπής. Βρισκόμαστε στην Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτού και όχι στην Επιτροπή ε, βιομηχανική Πολιτικής, ούτε στην Επιτροπή Απασχόλησης εδώ μέσα. Και γι' αυτό πάνω απ' όλα θα πρέπει να μεριμνούμε για την προστασία του καταναλωτή όχι να επιδιώκουμε άλλους στόχους. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσδορίζουμε εμείς ως ομάδα ως πάγια τακτική. Θεωρώ ότι η κυρία Σαρτόρ είναι μια καλή εισηγήτρια, έχει επισημάνει τα σημαντικότερα σημεία, την υποστηρίζουμε και περιμένουμε να δούμε στην πράξη. Δεν έχω μπορέσει να κοιτάξω ε, στις λεπτομέρειές της την έκθεση, αλλά θα το ε, πράξω φυσικά το ταχύτερο δυνατό και θα την υποστηρίξουμε στην προσπάθειά της. Κύριε Φόξ, ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον κύριο Κρότσμαν για τα σχόλιά του, γιατί συμφωνώ πολύ με όλα όσα είπε. Ιδιαίτερο να πω ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα φτάσει τίποτε στην αγορά ω προϊόν που θα μπορούσε να βλάψει τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Στη μελέτη εντεκτύπου σημείωσα κατά την παρουσίαση ότι οι νέοι κανόνε θα μειώσουν τι δοκιμέ σε ζώα. Αυτό το καλωσορίζουμε θερμά ως εξέλιξη. Επίσης η εξοικονόμηση που προτείνεται από τη μελέτη που είναι πολύ σημαντική. Η μείωση των τιμών θα ωφελήσει τους καταναλωτές. Όπως και η μείωση του κόστους μπορεί να προωθήσει και να δώσει μεγαλύτερη όθηση στην έρευνα και την κοινοτομία. Θα συμφωνήσω και με τα σχόλια της σοσιαλιστού συναδέλφου που μίλησε για μεγαλύτερη προστασία. Δεν ε, μπορώ παρά να συμφωνήσω. Και τις ανησυχίες της κυρίας Κλάσης μερίζομαι για το τι είναι και τι δεν είναι χαμηλού κινδύνου προϊόν. Θα ήθελα έναν ορισμό για, το χαμηλού, για τις ουσίες χαμηλού κινδύνου. Να διευρυνθεί ο ορισμός και να, να ελέγχονται περισσότερες ουσίες μέσα από το κεντρικό μας σύστημα. Ένα σύστημα που θα μειώνει τις τιμές και θα ωφελεί τους καταναλωτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριο Μπαρνιέ, η κυρία Σάλντε και η κυρία Γκέπχαρτ θέλει να δευτερολογήσει. Όμω να έχουμε το χρόνο για να έχουν το λόγο να τοποθετηθούν, το χρόνο να τοποθετηθούν και η Επιτροπή και η κυρία Σαρτόρη ξανά. Κύριε Μπαρνιέ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε σε μια συζήτηση για την αποτίμηση τη στρατηγική που προτείνεται από την Επιτροπή. Του γενικού προσανατολισμού κοιτάζουμε για να ετοιμάσουμε σωστά τις επόμενες φάσεις εξέτασης ενός κειμένου που εγώ θεωρώ άκρο σημαντικό, όπως και άλλα θεμελιώδη κείμενα που σήμερα εξετάσαμε. Και άλλα παρόμοια κείμενα από τα προηγούμενα χρόνια με την ευθεία και τη συνδρομή του Κοινοβουλίου ετοιμάσαμε. Το πρώτο ερώτημα που έχω να θέσω προς την Επιτροπή και θα με επιτρέψετε, Πρόεδρε, να βιαστώ λιγάκι γιατί υπάρχουν και τα προβλήματα με του υδροδρόμους σήμερα που μα ε, επιβάλλουν περαιτέρω φραγμούς αλλά πρέπει να θέσω το ερώτημα αυτό προ την Επιτροπή και να περιμένω και την απάντησή τη. Η παρουσία σα ήταν ιδιαίτερα σαφή και ολοκληρωμένη κυρία μου αλλά πού έχουμε φτάσει με το πακέτο για τα ζυζανιοκτώνα. Είναι ένα πακέτο το οποίο το θυμάμαι από προηγούμενα χρόνια εγκρίθηκε και η Γαλλική Προεδρία και εγώ είχαμε συνεργαστεί στενά για την έγκρισή του. Πώς αξιολογείτε την ε, παρακολούθηση των μέτρων αυτών και την υλοποίησή τους. Γιατί τα ζυζανιοκτώνα όπως και τα διοκτώνα είναι προϊόντα που κατά την άποψή μου είμαι ότι μπορούμε να πετύχουμε εξοικονόμηση. Ακόμα και αν αυτό δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στις επιχειρήσεις προς στιγμή. Ή αν πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι παντού τα κείμενα, θα πρέπει, τα οι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και θα πρέπει να σκεφτούμε και κατά πόσο τα εμπόδια αυτά μπορεί να αφορούν και την ανθρώπινη υγεία ή όχι. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Στην Επιτροπή εδώ το θέμα προτεραιότητας και όλα τα άλλα έπονται είναι εάν μπορούμε να δεχτούμε τους ε, περαιτέρω φραγμούς για σκοπούς προάσπισης της ανθρώπινης υγείας και εφόσον δεν υπάρχει και στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της αγοράς ή άνηση μεταχείριση. Θέλω λοιπόν να ξέρω τι συμβαίνει με το πακέτο των ζυζανιοκτώνων, τι συμβαίνει με το ρίτς. Και βεβαίως με τους όρους ισότιμης και αυστηρής υλοποίησης των κανόνων αυτών σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ την κυρία Σαρτόρη και την κυρία Κλάς για τις παρατηρήσεις που έκαναν ιδίως για τα θέματα της έρευνας, όπου σαφώς θα επιτελεστεί πρόοδος αν πετύχουμε εξοικονόμηση κονδυλίων. Και για τη συνέχεια των εργασιών μας, σημαντικό νομίζω θα είναι να γνωρίζουμε, όπως ρώτησε η κυρία Κλάς και πολλοί το ανέφεραν, όπως και εσείς οι ίδια, για την εισαγωγή των προϊόντων από τρίτες χώρες. Τι θα γίνει με αυτά. Ό,τι εισάγεται, όπως είπε η κυρία Κλάς, για να αναφέρω κυριολεκτικά την παρέμβασή τη, θα πρέπει να σέβεται απολύτω του κοινοτικού κανόνε. Η Επιτροπή λοιπόν προβλέπει πρωτοβουλίε ή ανέλαβε πρωτοβουλίε για να εναρμονίσει, να ευνοήσει, να βελτιώσει την δημιουργία εθνικών υπηρεσιών που θα ασχολούνται ακριβώ με του ελέγχου στα σύνορα, του λιμένε ή του αερολιμένε τη Ευρώπη και για άλλα θέματα βεβαίως, όπως η προστασία των καταναλωτών της Ευρώπης για τα... στην περίπτωση των τροφίμων που εισάγονται. Αλλά και εδώ, στα διοκτώνα, είναι σημαντικό να ξέρουμε αν η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλίες, ώστε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, της εσωτερικής αυτής αγοράς, πρόκειται να ανταλλάξουν, να εξισορροπήσουν, να δημιουργήσουν ένα σύστημα εχνηλασιμότητας των προϊόντων. Είναι σημαντικό αυτό για τα προσεχή χρόνια. Να ξέρουμε που έχουμε φτάσει ως προς την εκπαίδευση και την ε, οργάνωση των εθνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τον έλεγχο των εισαγόμενων προϊόντων. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπανιέλη ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ εύστοχα αυτά που μας είπατε, ανάλογα με την πείρα σας. Κύριε Σαλντεμόζο, κύριε Γκέμπχαρτ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι για να μπορέσει να λάβει το λόγο η Κομισιόν, η κυρία Σατόρη και η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όχι, δεν πρόκειται να με μακρηγορήσω. Λέει η κυρία Σάλντε Βεβαίως και μας απασχολεί η ασφάλεια των καταναλωτών. Και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε κάποιες δαπάνες Τώρα έχω μια ερώτηση συγκεκριμένη προς την Επιτροπή. Ακούει, δεν ακούει, ποιος ξέρει. Είναι συγκεκριμένη ερώτηση που έχω να σας υποβάλω. Διότι αναφέρατε ότι είναι σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Τι γίνεται τώρα από πλευρά εποπτεία τη αγορά. Έγινε κάποια έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπιστώθηκε ότι δύο κράτη-μέλη αποφάσισαν να δαπανίσουν περισσότερα χρήματα όσον αφορά την τελειοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών. Άρα η εποπτεία απαιτεί περισσότερο χρήμα. Εάν απλουστεύσετε τις ισχύουσες διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη δουλειά με πλευράς υποπτίας. Είναι ρεαλιστικό όμως αυτό, εκτός από την δειγματοληψία. Μήπως μπορούμε με άλλο τρόπο να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να ε, ασχοληθούν πιο αποτελεσματικά με το θέμα. Πώς θα επιβληθεί η νομοθεσία. Και έχετε επίση και την εκθεσή σα που μα βοηθάει σε αυτό το θέμα. Κυρία Γκέμπχαρτ, παρακαλώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φόξ, να ακούτε πιο προσεκτικό όταν μιλάω. Ιδιαίτερα εσείς. Δεν είπα ότι θέλω περισσότερη γραφειοκρατία. Είπα ότι πρέπει να προσέξουμε με την από διάρθρωση της γραφειοκρατίας, την απαλλαγή από τη γραφειοκρατία, να προσέξουμε να μην επιδεινωθεί το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τι είπατε κι εσείς, ότι εδώ δεν έχουμε, δεν είμαστε, και υπόθηκε μάλλον και από άλλοι συνάδελφοι, ότι δεν είμαστε εδώ στην Επιτροπή Βιομηχανίας, αλλά στην Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή. Και χαιρετίζω τα όσα είπε Σορτόρη για το τι πρέπει να επαληθεύσουμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπόθεση αυτή. Ναι, ίσως να λάβατε κι εσείς αυτή την ανακοίνωση τύπου, από αυτή τη γερμανική οργάνωση που έχω λάβει κι εγώ, ε, αλλά τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Συγκεκριμενοποιώντας τη δουλειά μας, βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα, ζητούμε από την Επιτροπή απαντήσεις και να δούμε, για να δούμε εάν ευσταθούν ή όχι οι ανησυχίες και οι φόβοι. Αυτό κάνουμε λοιπόν. Δεν αρχίζουμε καταγγελίες άκριτες λέγοντας είπε μία οργάνωση κτλ. Όχι. Ελέγχουμε και μετά. Θα συνεχιστεί η συζήτηση οπωσδήποτε, αλλά για ακούσουμε στο δεκάλεπτο που μένει τους συζητητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Mr. President. Επιτροπή. Σιγά σιγά βρίσκεται το όνομά μου, το μαθαίνετε στην επόμενη συνάντηση θα το πείτε τέλεια. Ευχαριστώ την κυρία Σατόρη, αλλά ευχαριστώ και τους άλλους ανθρώπους της Επιτροπής σα, Διότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητικά τόσα είπαν για την πρότασή μας. Συγχωρήστε μας πρώτα πρώτα, διότι δεν έγινε η παρουσίαση όπως θα θέλατε της ε, περίληψης της ε, μελέτης επιπτώσεων. Πολλές φορές δεν μπορούμε να μαντέψουμε τι θέλει ο αποδέκτης του έργου μας. Πάντως, το αποτέλεσμα της ε, μελέτης επιπτώσεων είναι στρατηγική σημασία και θα επανέλθω σε αυτό. Επίσης, Θέλω να σας τονίσω ξεκάθαρα ότι ο στόχος της πρότασης μας με τίποτα δεν είναι να μειώσουμε το, το, το, το επίπεδο, να κατεβάσουμε τον πύχη όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η πρόταση είναι ότι Έχουμε ήδη κάποιε διατάξει, έχουμε τέτοια όρθα συνθήκε, αλλά δεν ε, είναι τόσο αποτελεσματική η διαδικασία αυτή, γιατί δεν είναι αποτελεσματική η συνοδευτική διαδικασία. Άρα, α βάλουμε μερικέ ακόμα διατάξει που θα βελτιώσουν την προσέγγιση του περιβάλλοντο. Πάρα πολύ σαφή κριτήρια αποκλεισμού. Να μην επιτρέπουμε τα πηγαίνοντα προϊόντα, καλά, καλά, μην πω στι λεπτομέρειε. Όμω, είναι σαφέ ότι αυτό είναι ο στόχο. Να βελτιωθεί και όχι να επιδεινωθεί η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα γίνει με ένα αποτελεσματικό σύστημα. Αυτό θα βοηθήσει τις ΜΜΕ, αλλά και τις άλλες εταιρείε να ενθαρρυνθούν και στο μέλλον να θέτουν σε εμπορία λιγότερα και λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. Έχουμε τα διοκτώνα, έχουμε χιλιάδες άλλες ουσίες και πολλές από αυτές χρησιμεύουν ως υποκατάστατα. Οπότε θα πρέπει να κάτσουν και να βρουν, αφού είναι δυνατόν, ποιε είναι υποκατάστατε ουσίε αντί για τι επικίνδυνε. Α γίνει σύγκριση και αν έχουμε ένα διοκτόνο που έχει κάποια ουσία που μπορεί να αντικατασταθεί, θα πρέπει να γίνει η σύγκριση με άλλα προϊόντα που είναι λιγότερο επικίνδυνο τρόπο να το κόστος Θέλουμε να μειωθεί το κόστος και ελέγχει ότι η κεντρική διαδικασία θα πρέπει να καλύψει περισσότερα. Τότε όμως θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά. 27-29 κρατημέλη θέλουμε να καλύψουμε. Και βέβαια ε, είναι πιο αποτελεσματικό από κάθε άλλη μέθοδο, διότι έτσι αν πάει κανείς σε μια διαδικασία καλύπτει όλη την αγορά θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο κοινωνικός φορέας μπορεί, έχει τους πόρους για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί στην πράξη. Άρα χρειάζεται μια προσέγγιση βαθμιδών. Πολύ σημαντικό αυτό. και να δούμε αν είναι αποτελεσματική η κεντρική διαδικασία που είναι στατική σημασία. Άρα να διαπιστώσουμε ότι θα λειτουργεί το κέντρο κατευθυνόμενο σύστημα ε, αντί για το σημερινό σύστημα σε εθνικό επίπεδο. Γιατί είδαμε τι γίνεται με τα παρασυτοκτόνα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι να υπάρχει ψηλό επίπεδο προστασία, αλλά να στο επίπεδο, στο επίπεδο παντού. Και να μην δεχτούμε να κατέβει ο πύχη λόγω της αμοιβία αναγνώριση. Να. Βλέπετε αυτά εδώ τα μαντιλάκια τα απολυμαντικά, υπάρχει παντού αυτό το προϊόν, να είμαστε σίγουροι ότι είναι αποτελεσματικό και θα πρέπει η απολύμανση να μην διαφέρει από το ένα κράτο στο άλλο. Ίσως υπάρχει ένα δικό πρόβλημα, να υπάρχει κάποιο είδους ε, ε, λοιμός σε κάποιο, σε κάποιο κράτος, αλλά για ποιο λόγο να μην έχουμε αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση. Να μην υπάρχει φραγμός. Και αν υπάρχει φραγμός από κάποιο κράτος μέλος, να παρέχεται επαρκής αιτιολόγηση. Να υπάρχει προστασία αλλά και να υπάρχει και λιγότερη γραφειοκρατία. Άκουσα κάτι για τα έχουν τα επεξεργασία, προϊόντα, για την ετικετοθεσία. Αλλά χρειάζεται αυτό για την ενεχνευσιμότητα. Πού να ξέρετε αν ο καναπές που πήρατε, αν έχει υποστεί κάποια επεξεργασία με χημικά, αν δεν υπάρχει η ετικετοθεσία. Άρα για την ενεχνευσιμότητα χρειάζεται. Φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει και αναφορά συγκεκριμένη στην έγκριση. Είναι και θέμα ανταγωνισμού. Το ανέφερε κάποιος βουλευτής γιατί στην ε, Ευρώπη όλοι οι παραγωγοί υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν μόνο εγκεκριμένε ε, ουσίες και υλικά. Τι γίνεται όμως με τα εισαγόμενα. είναι πιο φτηνά, δεν έχουν υποστεί τέτοιε διαδικασίε έγκριση. Και επομένω χρειάζεται η ετικέτα. Βέβαια, όπω για κάθε νέο νομοθέτημα, χρειάζεται να υπάρχει και επιβολή και εφαρμογή του νόμου. Και ταυτόχρονα να βοηθούμε τα τελωνία να είναι ενημερωμένα όπως ε, για την ασφάλεια των παιχνιδιών, όπως γίνεται για κάθε έλεγχο στα σύνορα της ε, Ένωσης, επομένως, να γνωρίζουν ενημερωμένοι όσο γίνεται περισσότεροι. Και στην ΕΚΑ υπάρχει ένα φόρο που αφορά τη συνεργασία αυτών των αργών. Βλέπω διπλωματικά και με τρόπο μου λέει ότι πρέπει να κλείσω. Πάντως νομίζουμε ότι είναι ισορροπημένη αυτή η ρύθμιση του κανονισμού. Προστασία του περιβάλλοντος αλλά και μείωση του κόστους. Και είμαστε πεπισμένοι ότι θα πάει καλά. Ο Πρόεδρος! Σας ευχαριστούμε. Πολύ χρήσιμο όσα είπατε. Κύριε Σαρτόρη, για να κλείσει. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο για το χρονοδιάγραμμα, κάτι άλλο. Ε, κάνα δύο λεπτά έχετε πριν. Τελειώσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω όλοι είμαστε ικανοποιημένοι από την σημερινή συζήτηση εδώ. Γιατί για όλους κατέστη σαφές τι μας περιμένει τι έχουμε να περιμένουμε από την εξέλιξη αυτού του κανονισμού και ποιος είναι επιδιωκόμενος σκοπός. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συμβολή τους. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προς στιγμή στα χέρια μας προβλέπει δεύτερη ανταλλαγή απόψεων στις 25-26 Ιανουαρίου. Ε, λήξη για την, ε, της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών 2 Φεβρουαρίου. Θεώρηση του σχεδίου γνωμοδότησης 23 Φεβρουαρίου 26 Φεβρουαρίου, όπως είπα, λήξη για την υποβολή, για την υποβολή τροπολογιών. 16 Μαρτίου εξέταση του κειμένου με τις τροπολογίες. Ψηφοφορίες στην ΙΜΚΟ 16, 17 Μαρτίου και 6-7 Απριλίου η ψηφοφορία. Και το Μάιο η τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι είναι αρκετό ο χρόνο που έχουμε μπροστά μα, όπω ζήτησαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, και σε συνεργασία με, τις, με τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ελπίζουμε και στη συνεργασία της Επιτροπής και ότι οι στόχοι που εκφράστηκαν ως επιδιωκόμενοι από πολλούς συναδέλφους θα τύχουν ευνοϊκής απόκρισης. Well, Σας ευχαριστούμε κυρία Σαρτόρη που ξεκαθαρίσατε και αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως έλεγα, τα έγγραφα μελέτης αντικτύπου διατίθενται από τη Γραμματεία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα να τα δείτε για να καταλάβετε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ πέρα. Εάν συμφωνούμε με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή καλύτερη προστασία των καταναλωτών και θελήσουμε να συσφίξουμε να κάνουμε πιο αυστηρούς μάλλον τους κανόνες για την εισαγωγή κανόνων και να βελτιώσουμε και τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υποθέτω ότι μια τέτοια προσέγγιση θα ικανοποιήσει όλα τα μέλη της Επιτροπής μας καθώς και τους καταναλωτές. Καθήκον μας λοιπόν είναι όλοι μαζί να επιδιώξουμε αυτό το είδους την ισορροπία η οποία είναι πάντοτε επιθυμητή σε κάθε πρόταση. Αυτό που θα συζητήσουμε μαζί Λοιπόν, είναι ακριβώ αυτά τα ζητήματα μαζί με εσά και του υπευθύνου του ντοσιέ. Επόμενη συνεδρίαση 16 Νοεμβρίου